Καλημέρα. Ας ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα λοιπόν Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το νούμερο 6. προς μια νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη 2011-2020. Η κυρία Κολόνσκα Μπομπίνσκα είναι αρμόδια. Θα της δώσω λοιπόν το λόγο. Θα γίνει μια συζήτηση. Ξέρετε πως 10 η ώρα ξεκινάνε οι ψηφοφορίες. Κυρία κολέσκα Μπομπίνσκα λοιπόν έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ακούσω στο δυνατόν περισσότερα σχόλια στην αρχική συζήτηση, οπότε δεν θα μακρηγορήσω. Η έκθεση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για να προετοιμάσει η Κομισιόν την ενεργειακή στρατηγική της για την Ευρώπη 2020. Έχει συμβουλευτικό δηλαδή χαρακτήρα. Γίνονται αυτή τη στιγμή διαβουλεύσεις με τους ε, κοινωνικούς εταίρους, διαφορέ οργανώσεις και κατά κάποιον τρόπο είναι μέρος αυτών των διαβουλεύσεων και αυτή η έκθεση. Γι' αυτό είναι σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ορίσει τους βασικούς στόχους ε, της ε, βασικής ενεργειακής στρατηγικής για τα επόμενα δέκα χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν να επικεντρωθώ στα ζητήματα κλειδιά και επειδή υπάρχουν αρκετά τέτοια θέματα. Πρέπει να επιλέξουμε προτεραιότητες, οπότε, έτσι ώστε η έκθεσή μας να μην γίνει σαν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο πάνω στο οποίο κρεμάμε τα πάντα ή σαν μια σούπα, αν και το γκούλας μου αρέσει εμένα. Εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει να ξεχνάμε το σημαντικότερο πράγμα εδώ πέρα, τις σημαντικότερες κατευθύνσεις που πρέπει να δώσουμε. Το δυσκολότερο πράγμα λοιπόν στη δουλειά μας είναι το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε. Η τελική εκδοχή αυτής της έκθεσης πρέπει να σταλεί στις 14 ε, Εβδόμου για μετάφραση και θα ψηφιστεί στην Επιτροπή μας ε, τον Σεπτέμβριο και μετά τον Οκτώβριο στο Στρασβούργο. Δεν υπάρχει λοιπόν αρκετός χρόνος για να προσπαθήσουμε να συνεννοηθούμε με άλλες επιτροπές ε, και ομάδες. Ο χρόνος πιέζει. Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό αποτελεσματικά, γι' αυτό και ζητάω τα σχόλιά σας ε, να γίνουν όσο δυνατόν πιο γρήγορα, είναι να γίνει γραπτός. Θα ήθελα να ζητήσω ειδικά από τους κοιόδεις ε, εισηγητές να στείλουν τα σχολιά τους το συντομότερο δυνατόν. Πρέπει να βρούμε έναν συμβιβασμό και να συντάξουμε μια καλή έκθεση, κάτι το οποίο βεβαίω δεν θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα επαναλαμβάνουμε κάποια πράγματα της ε, Ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη, πράγματα σημαντικά τα οποία θα συζητηθούν από μας και η βασική ιδέα στην ε, έκθεση αυτή είναι η ευρωπαϊκή στόχη στην ενεργειακή πολιτική, να εγγυηθούμε την ε, ασφαλή και σταθερή πρόσβαση στην ενέργεια με σταθερές τιμές για τους οικιακούς και επαγγελματικούς καταναλωτές. Ε, να εξοικονομήσουμε βεβαίω και ενέργεια και να προωθηθεί η καινοτομία και να μειωθούν οι κομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό το οποίο αξίζει να τονίσουμε είναι πως η Κομισιόν στην εκθεσή της, ε, και αυτό τονίζουμε πάνω απ' όλα, θέλει να διασφαλίσει πως ε, θα συμμορφωθούμε με όλες τις υποχρεώσεις που έχουμε τονίζεται δε στην έκθεση για πρώτη φορά πώς θα πρέπει να εφαρμοστούν οι κανόνες και υπάρχουν και κυρώσεις για την ε, μη συμμόρφωση. Και μάλιστα λέγεται πως ε, αναφέρεται πως ε, κάποιες γενικές διευθύνσεις θα χρησιμοποιήσουν κάποιες, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαδικασία παραβάση. Αυτά είναι τα σημεία στα οποία έχουμε συμφωνήσει. Δεύτερον, η ημερομηνία εφαρμογή. βεβαίω είναι η 3η Μαρτίου του επόμενου έτους. Οπότε υπάρχουν ήδη κάποια πράγματα. Και η Κομισιόν φανταζομαι θα προετοιμάσει ήδη κάποια έγγραφα για τη διαδικασία αυτή η παραβάση. Αμέσως μετά φαντάζομαι την προθεσμία του Μαρτίου και όχι μόνο θα πρέπει να συμμορφωθούν με διάφορες προδιαγραφές στα κράτη-μέλη, αλλά και με Θα όσα αναφέρω σε διεθνείς συμφωνίες και στα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τονίζεται εδώ πέρα επίσης πάρα πολύ η υποδομή, το ζήτημα της υποδομής. Τονίζω πως οι στόχοι αυτοί είναι οι γνωστοί στόχοι που έχουμε στην ευρωπαϊκή στρατηγική, γενική αυτή η στόχη, αλλά τονίζεται πως θα πρέπει να δούμε κάποια πράγματα διαφορετικά από ό,τι κάναμε μέχρι στιγμής. Θα ήθελα τώρα να αναφέρω την υποδομή. Έχουμε λοιπόν τους στόχους αυτούς για το 2000. 20, αλλά μόνο συζητήσει θα έχουμε εάν δεν έχουμε έξυπνα δίκτυα. Είναι σαφές από την έκθεση πώς θα πρέπει, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καλύψουμε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με έξυπνα δίκτυα και να προχωρήσουμε και πέρα από τα σύνορα των κρατών μελών και πέρα από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε τα δίκτυα αυτά να συμπεριλάβουν και άλλες χώρες. Λεφτά τώρα, αν θα μας δώσουν ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Χρειαζόμαστε εκατομμύρια ευρώ για αυτές τις υποδομές και η έκθεση υπογραμμίζει ιδιαίτερα την χρήση των μηχανισμών της αγοράς και επομένως θα πρέπει να εξετάσουμε αν μέσα από του μηχανισμού τη αγορά μπορούμε να βρούμε αρκετά χρήματα για να καλυφθεί το κόστο των υποδομών. Στην έκθεση επίση αναφέρεται το δυναμικό το οποίο υπάρχει για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας, αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας και εδώ μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη διασαφήνιση και είναι μεγάλη σημασία επίσης όπως αναφέρεται στην έκθεση η εξωτερική διάσταση της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή θα πρέπει να διαμορφώσει μια πολιτική κοινή στον τομέα αυτό και θα ήθελα από κοινού όλοι οι συνάδελφοι να αποσαφηνίσουμε τελείως τις ε, βασικές πτυχές της εξωτερικής μας πολιτικής για τα θέματα ενέργειας, επίσης την ανάπτυξη διασυνδέσεων και διευρωπαϊκών δικτύων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ποιο τρόπο θα πρέπει να πραγματοποιηθούν αυτά, αν θα χρειαστεί ένα ειδικό είδος συμβάσεων, πώ θα επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες. Τίποτα από όλα αυτά δεν αναφέρεται αρκετά εκπεφρασμένα στην έκθεση αυτή. Χρειάζεται να δώσουμε και κάποιες δικές μας ιδέες για να τη βελτιώσουμε λοιπόν. Και εν τέλει, η έκθεση υπογραμμίζει τη σημασία της έρευνας και το σχέδιο αυτό είναι ένα σημαντικό συστατικό της συνολικής μας δράσης για τη μείωση του διοξιδίου, των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τα κύρια στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στο ερευνητικό αυτό σχέδιο και επιπλέον υπάρχει ένας ακόμα χώρος στον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να σκεφτούμε και τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μια περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας που χρησιμοποιούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μειώσουμε και την εξάρτησή μας από εξωτερικές Ευρωπαϊκής Ένωσης πηγές ενέργειας. Αξίζει τον κόπο να κάνουμε προσπάθειες και ερεύνα προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης η έκθεση δεν λέγονται αρκετά για την εφαρμογή του άρθρου 194 της Συνδίκης Λισαβόνας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού και επίσης η έννοια της αλληλεγγύης που ανέφερε ο Επίτροπος κ. Τιγκέρ αναφέρεται σποραδικά μονάχα στην έκθεση χωρίς όμως αρκετή υπογράμμιση. Πρέπει να τονίσουμε ότι η ασφάλεια εφοδιασμού είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να τονιστεί όπως και η αλληλεγγύη. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, αν δούμε ποια είναι η διαμάχη η οποία αναδύεται συνέχεια και μετά εξαφανίζεται μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας. Δεν ξέρουμε πότε θα ξανααναδυθεί αυτή η σύγκρουση, αλλά θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας αυτή τη δυνατότητα. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τη βοήθεια όλων των μελών της Επιτροπής που με ακούσατε και όλες. Θα σας ευχαριστήσω, λέει και ο Πρόεδρος, για την παρουσίασή σας. Οι σκιώδεις τώρα έχουν το λόγο. Κυρία Μεσάρους. Κύριος Μεσάρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έργο της, γιατί αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για μας. Μετά από την κύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διαφορετικό τρόπο. Θα είναι και τμήμα της εντολής μας, μαζί με τα κράτη-μέλη, να θεσπίσουμε μια νέα πολιτική. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ενεργειακή ασφάλεια, να προωθήσουμε την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας, ιδίως να αναπτύξουμε περαιτέρω τη χρήση των ανανεωσίμων ενεργειών και θέλουμε φυσικά να υπάρξει και καλύτερη διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον τρόπο αυτό τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν <clears throat> τους πόρους οι οποίοι είναι καταλληλότεροι για τα κράτη-μέλη αυτά και να μπορούν να καθορίσουν την ενεργειακή διάρθρωση της, του εφοδιασμού τους σε ενέργεια. Η περαιτέρω λοιπόν ανάπτυξη αυτών των ε, των αναγκών σε ενέργεια σημαίνει και μεγαλύτερη ανάγκη διαδικτύωση στον ενεργειακό τομέα. Το 2030 το 65% της, ε, των αναγκών της ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εισάγονται από τρίτες χώρες. 80% στην περίπτωση του φυσικού αερίου. Ως εκ τούτου πρέπει να εξασφαλίσουμε την ε, παρουσία διαφοροποιημένων πηγών ενέργειας και των καταλήλων διαδρόμων ενεργείας. <clears throat> Οι σταθμοί ενέργειας έχουν περιορισμένο χρόνο ζωής και πρέπει να αντικαθίστανται περιοδικά. Χρειαζόμαστε χρήματα της τάξης των 100 δισεκατομμύριων ευρώ για την κατασκευή νέων σταθμών και την διάλυση των προηγουμένων σταθμών ενέργειας με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι οικολογικά ασφαλής. Πρέπει να εξασφαλίσουμε επίσης τη συντήρηση των προηγουμένων σταθμών και να ξαναθέσουμε επιτάπητος το θέμα της πυρηνικής ενέργειας. Υπάρχουν και νέες ιδέες όπως η θερμοπυρηνική σύνδεξη, όπως παραδείγματο χάρη το σχέδιο ΙΤΕΡ. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς να εξασφαλίσει πιο καθαρή ενέργεια στο μέλλον. Θέλουμε λοιπόν να τονίσουμε τις, τους τρεις αυτούς πυλώνες, αποδοτική χρήση ενέργειας, μείωση των απολειών ενέργειας και μεγαλύτερη αλληλεγγύη στα θέματα της ενέργειας. Όλα αυτά σημαίνουν ότι πρέπει να τροποποιήσουμε τις μεθόδους μα. Αυτό δεν μπορεί να είναι μια διαδικασία που θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να επιτύχουμε τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς ενέργειας, μειώνων έτσι το ρόλο των εθνικών κρατών, αλλά ενισχύοντα συγχρόνω και το ρόλο των περιφερειών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τι χώρε τη Κεντροανατολική Ευρώπη, όπου η περιφερειακή συνεργασία είναι στα γενοφάσκια Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Γκίρεκ, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όταν μιλάμε για ενεργειακά ζητήματα πρέπει πάντα να θυμόμαστε το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Η ενέργεια και η ανταγωνιστικότητα είναι απολύτως ε, συνδεδεμένες. Από την άλλη, κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετικό ενεργειακό μείγμα. Οπότε η ανταγωνιστικότητα του κάθε κράτους μέλους ε, δεν είναι ίδια. Όμως αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη καθώς υπάρχει εδώ πέρα μία ενιαία προσέγγιση στην ε, ενεργειακή στρατηγική. Δεν μπορούμε να αναρμονίσουμε τις πηγές ενέργειας. Δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε μία μέση λύση. Μία τέτοια προσπάθεια ε, τέτοια οδήγησε στο πακέτο του κλίματος και θυμάμαι πως ε, το πακέτο αυτό προετοιμάστηκε έχοντας ε, κατά νου την 15η ε, σύνοδο των συμβαλωμένων μερών στην Κοπενχάγη κάτι το οποίο τελικά δεν ήταν ρεαλιστικό γιατί το σκεπτικό ήταν ότι θα πείσουμε εμείς τον κόσμο να μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα αλλά τώρα εκ των υστέρων ξέρουμε ποιο ήταν τα, τα αποτελέσματα στην Κοπενχάγη. Εάν επιμείνουμε λοιπόν σε αυτές τις ε, διατάξεις η Ευρώπη δεν θα είναι πλέον ανταγωνιστική. Μπορούμε να μιλάμε για την Ευρώπη του 2020, για τη στρατηγική, για το τι θέλουμε να πετύχουμε, αλλά όλα αυτά θα παραμείνουν ε, όνειρο απατηλός αντί Λισαβόνα και κάπως έτσι μη ρεαλιστικό. Οπότε πρέπει να επανεξετάσουμε αυτό το πακέτο το κλιματικό, πρέπει να επικεντρωθούμε στα ρεαλιστικά του στοιχεία και εδώ πέρα εννοώ την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας είναι και πρέπει να είναι η βάση της ανάπτυξης ε, του ενεργειακού τομέα. Επιπλέον η Ευρώπη είναι διχασμένη όσον αφορά την ατομική ενέργεια. Γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί δεν μπορούμε στην έκθεση αυτή να έχουμε κάποιες διατάξεις οι οποίες ε, θα μας δώσουν ε, μία νέα ευκαιρία για την πυρηνική ενέργεια στην Ευρώπη. Χωρίς ε, κάτι τέτοιο δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Και επίσης υπάρχουν ε, κάποια σημεία που πρέπει να δεχτούμε, δηλαδή δίκτυα χαμηλής ποιότητας, έλλειψη διασυνδέσεων που αναφέρθηκε ήδη στην έκθεση. Και το λεγόμενο φαινόμενο Κάρινγκτον, δεν ξέρω αν το ξέρετε όλοι. Ε, δεν ξέρω αν ε, το έχετε ακούσει και με συγχωρείτε, θα, θα σας δώσω ορισμένες πληροφορίες. Στον 19ο αιώνα τα δίκτυα τηλεπικοινωνίας είχαν προβλήματα λόγω της ε, ηλεκτρομαγνητικής ε, εκνοβολίας του ηλίου. Δεν υπήρχαν πάρα πολλά δίκτυα και τι συνέβαινε καίγονταν οι μετασχηματιστές. Τι θα συνέβαινε τώρα εάν είχαμε μια αύξηση της ηλεκτρομαγνητικής ακνοβολίας του ηλίου. Τώρα που έχουμε τόσους πολλούς ε, μετασχηματιστές, τόσες διασυνδέσεις στα δίκτυα, αν αντιμετωπίσουμε ένα blackout σε μια μεγάλη περιοχή του κόσμου. Αυτά δεν είναι επιστημονική φαντασία που σας λέω είναι κάτι το πιθανό. Οι σχεδιαστές πρέπει να τα λάβουν αυτά υπόψη. Οι Αμερικάνοι ήδη το κάνουν. Οπότε θα ήθελα να τονίσω αυτό το σημείο σημαντικό στην ε, παρέμβασή μου. Πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε το ενεργειακό πακέτο. Οι στόχοι του ήταν υπερβολικά φιλόδοξη και η προσέγγιση ήταν μια έτσι μέση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σιμάνσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε με έγγραφα αυτού του χαρακτήρα, τα οποία περιλαμβάνουν τον όρο στρατηγική στον τίτλο τους είναι η εξισορρόπηση των διαφόρων στόχων και προσπαθειών. Ίσως δεν είναι τόσο δύσκολο να καταρτήσει κανείς ένα κατάλογο όλων των ετοιμάτων που έχουμε, τα οποία μπορούν να διατυπωθούν από τα μέλη της Επιτροπής μας. <clears throat> Μιλάμε για ένα σενάριο το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί σε βάθος χρόνου. Και στο προηγούμενο σχέδιο δράση είχαμε δύο κατηγορίες ετοιμάτων. Καταρχήν, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ήταν η πρώτη κατηγορία και η δεύτερη κατηγορία είχε να κάνει με θέματα εφοδιασμού σε ενέργεια. Αλλά τα δύο αυτά ζητήματα είναι αλληλένδετα και συνδέονται μεταξύ τους. Η αποδοτικότητα της ενέργειας, η χρήση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας ενισχύουν και την ασφάλεια εφοδιασμού. Όλα αυτά θα χρειαστούν χρόνο φυσικά. Αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας δεν επαρκούν για να μπορέσουμε να εξαλείψουμε μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα όλες τις πηγές παραγωγής ενέργειας που εκπέμπουν αερία θερμοκηπίου. Στην κεντροανατολική Ευρώπη βλέπετε πραγματικά να υπάρχει μία σύγκρουση μεταξύ στόχων ασφάλειας εφοδιασμού και προστασίας του κλίματος και αυτή η έλλειψη ισορροπίας και η σύγκρουση κατευθύνσεων μπορεί να οδηγήσει ακόμα μεγαλύτερη εξάρτηση από το φυσικό αέριο, επομένως και ακόμα πιο σοβαρά προβλήματα ασφάλειας εφοδιασμού. Και εδώ φυσικά εμπλέκονται και οι εταιρείε οι οποίες εισάγουν ενέργεια από τη Ρωσία, η ενδιάμεση. Ο ρόλος τους είναι πάρα πολύ σημαντικός σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού σε ενέργεια, ιδίως για την Ανατολική Ευρώπη. Δεν πρέπει λοιπόν να παραμείνουμε σε ένα επίπεδο απαρίθμησης όλων των ετοιμάτων μας. Θα πρέπει να εστιάσουμε καλύτερα στο πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με καλύτερο τρόπο όλα αυτά τα θέματα Καταρχήν πρέπει να εγγυηθούμε σωστές υποδομές, χωρίς να αποκλείουμε το πιο πολιτικό, την πιο πολιτική πτυχή του θέματος. Thank you, uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Τούρμ. Υπάρχει δυνατότητα να αποκτήσει πιο στρατηγικό χαρακτήρα αυτό το έγγραφο. Όταν ε, τελείωσα, όταν το διάβασα, σκέφτηκα... Εντάξει, καλές όλες αυτές οι ιδέες, αλλά μου φάνηκε σαν ένα συνοθήλευμα ιδεών. Μου φάνηκε ότι δεν υπήρχε μια σωστή ιεράρχηση των ιδεών. Δεν υπήρχε κάποια σωστή σειρά. Για τις ανταγωνιστικές τιμές. Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας το 95% της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου που πωλείται στην Ευρώπη πωλείται από 12 μόνο εταιρείες. Η υλοποίηση λοιπόν του τρίτου πακέτου, η ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των, αρχών ανταγωνισμού και της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στις Βρυξέλλες ε, πρέπει να καταπολεμήσουν αυτή την ανάπτυξη των ολιγοπολιακών καταστάσεων στην Ευρώπη. Βασικά το Γαλλικό Κοινοβούλιο αυτές τις μέρες ενσωματώνει στο Εθνικό Δίκαιο το δεύτερο πακέτο της ενέργειας και έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε τη διάρθρωση της γαλλικής αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Οι γαλλικές εταιρείες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι πολύ δραστήριες και παρούσες στη Βρετανική αγορά, στην Ισπανική αγορά. Η ΕΟΝ με 2,5% μερίδιο αγοράς και το Γαλλικό Κοινοβούλιο δεν δεν προσπαθεί να προστατεύσει τις δικές του εταιρείες. Προσπαθεί να, συγγνώμη, να προστατεύσει τις δικές του εταιρείες και την ε, θέση τους ε, εντός της Γαλλίας αλλά και εντός της Ευρώπης. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε προτεραιότητα το τομέα αυτό. Δεύτερον, κάτι άλλο που πρέπει να καταλάβουμε επίσης. Η ενέργεια είναι ένας κυκλικός επιχειρηματικός κλάδος τα τελευταία 40-45 χρόνια. Είναι πολύ φτηνή η ηλεκτρική ενέργεια ανά κιλοβατόρα. Οι τιμές είναι πολύ χαμηλές. Ήταν πολύ χαμηλές, ιδίως στις αρχές της δεκαετίας του 90 και στις αρχές του της δεκαετίας του 2000. Όταν ε, ενοποιήθηκε κάπως η αγορά των 27 κρατών μελών υπήρχε μεγαλύτερη προσφορά παρά ζήτηση. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη επίγνωση ότι από τώρα μέχρι το 2025 θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τρεις βαθιές τάσεις. Ε, τρεις σημαντικές τάσεις. Το ίμιση, το 2 τρίτα όλου του ηλεκτρικού ρεύματος, όλων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη θα πρέπει να ανανεωθούν γιατί φτάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους, άρα θα αυξηθούν οι τιμές. Δεύτερον, η υποδομή διανομής επίσης φτάνει στο τέλος της ζωής της. Ακόμα και σε μια χώρα όπως η Γερμανία, αν δείτε τη δυτική, εντάξει, και στην Ανατολική Γερμανία χτίστηκαν πολύ καινούργιοι, πολλές καινούργιες εγκαταστάσεις διανομής, αλλά στη Δυτική Γερμανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη ε, οι γραμμές υψηλής τάσης ε, έχουν, κλείνουν έναν κύκλο ζωής 40, 45, 50 ετών και στην Ιταλία και στη Γαλλία. Οπότε τόσο η διανομή ε, όσο και η μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος είναι κάτι, ένας τομέας που θα ακριβίνει. Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος λοιπόν θα ανέβουν. Διαφορετικά δεν θα υπάρχουν κίνητρα για να ε, επεκτείνουν την υποδομή, να την ανανεώσουν οι επενδυτές. Ε, αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί ως την τιμή, πρέπει να δούμε και την άλλη παράμετρο, τον όγκο της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου που θα χρησιμοποιούμε. Ε, για να διατηρήσουμε το γενικό κόστος για την οικονομία σε εύλογα επίπεδα, θα πρέπει τα επόμενα χρόνια να ασχοληθούμε πολύ περισσότερο με την αποδοτική χρήση της ενέργειας, για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε αυτή την ισορροπία και να αναχαιτήσουμε αυτή την τάση ανόδου της ηλεκτρικής ενέργειας ανά Διαφορετικά οι οικονομικοί νόμοι θα επικρατήσουν σε αυτό το τόσο σημαντικό τομέα για την οικονομία. Ερχόμενος τώρα στην ασφάλεια. Ανησυχώ λίγο περισσότερο από άλλους συναδέλφους. Γιατί ε, η Gazprom και άλλες εταιρείες θα πρέπει να, να κάνουν υποχωρήσεις. Μετά από την Ουκρανική κρίση η κατάσταση έχει αλλάξει και χρειαζόμαστε ρευστό για τις επενδύσεις. Γι' αυτό υποχώρησαν. Και εμείς ως Ευρωπαίοι είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι σήμερα από ό,τι ήμασταν πριν από 20 χρόνια. Νομίζω ότι ε, οριστικοποιούμε τώρα τον κανονισμό για την ασφάλεια του ανεφοδιασμού σε φυσικό αέριο και οι ροές φυσικού αερίου στην Ευρώπη ε, θα χαρακτηριστεί από κρίσεις και από αναχέτηση της ροής. Το αέριο αποσβεστολιθικό σχιστόλιθο δεν ξέρω τι προοπτικές έχει στην Ευρώπη. Πρέπει να είμαστε πολύ επικεντρωμένοι. Πρέπει να παροτρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ερευνήσει πού υπάρχει αέριο ασβεστολιθικής φύσεως στην Ευρώπη νομίζω σε μέρη της ε, δημοκρατίας της Τσεχίας, ε, στην Κροατία, νομίζω στα, στην περιοχή των Βαλκανίων, γιατί αυτό θα μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική πηγή ανεφοδιασμού και άρα θα αυξήσει την ασφάλειά μας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ένα άλλο κεφάλαιο που διαθέτουμε για να μειώσουμε την εξάρτησή μας από, από την ενέργεια και αυτό το θέμα συνδέεται επίσης με την υποδομή. Νομίζω το πακέτο των υποδομών είναι ένα από τα θέματα κλειδιά που πρέπει να σχεδιαστούν πολύ προσεκτικά. Δύο πράγματα εδώ. Ένα για την ε, βιωσιμότητα των, ε, του δικτύου διανομής. Αν θέλουμε να έχουμε ένα βάρος και να μας ακούσουν οι χαράκτες, ε, πολιτικοί, πρέπει να οι χαράκτες πολιτικής, πρέπει να απομακρυνθούμε από την προσέγγιση του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Δεν μπορούμε να έχουμε έναν πολύ μικρό προϋπολογισμό για να χρηματοδοτήσουμε δεκάδες δίκτυα διανομής στην Ευρώπη. Αυτά είναι ψίχουλα. Εδώ μιλάμε για εκατοντάδες ε, εκατομμύρια, αν όχι δισεκατομμύρια επενδύσεων. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποιοι είναι οι πέντε ή έξι διάδρομοι όπου θα έχουμε τεράστιες ροές ε, ιδίω αιωλικής ενέργειας μετά το 2020. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτήσει πολύ αναλυτικά σενάρια για την κατάσταση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πέρα από τον ορίζοντα το 2020 γιατί πρέπει να προλάβουμε τις εξελίξεις. Και τέλος, κάτι που είναι πρέπει να προσέξουμε είναι τα οικονομικά. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τους πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων τραπεζών και τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και να δημιουργήσουμε εργαλεία που να δημιουργήσουν μόχλευση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί η αποδοτική χρήση της ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντική και για την ασφάλεια του ανεφοδιασμού και για την ε, διατήρηση των ανταγωνιστικών τιμών στο πακέτο της ενέργειας και νομίζω ότι πρέπει να τους δώσουμε μεγαλύτερη προτεραιότητα. Νομίζω ότι πρέπει να είναι υπαριθμόν ένα προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια. Έτσι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε πραγματικά την ενεργειακή μας πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τούρμες. Υπενθυμίζω πως έχουμε 24 λεπτά ακόμα. Έξι συνάδελφοι έχουν ζητήσει να λάβουν τον λόγο, συν η συγγήτρια συν η Κομισιόν. Αν συνεχίσουμε έτσι δεν θα προλάβουμε όλοι. Προτείνω να περιοριστούμε σε ένα-δύο λεπτά, αλλιώς δεν θα μπορέσουν να μιλήσουν όλοι και στις 10 η ώρα ψηφίζουμε. Ο κύριος Μπαλτσίτης κατόπιν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε δίκιο, πρέπει να είμαστε πιο σύντομοι για να μπορούν να μιλήσουν όλοι τελικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την παρουσίαση της ε, έκθεσής της. Ο τομέας της ενέργειας οπωσδήποτε θα παραμείνει ε, σε άμεση σχέση με την ανταγωνιστικότητα και των χωρών και της Ένωσης ε, στο σύνολό της. Οπότε δεν πρέπει να μιλάμε για ανταγωνισμό εντός της Ένωσης, αλλά για ανταγωνισμό με τις εξωτερικές αγορές. Αυτό έχει εξαιρετική σημασία. Θέλω να αναφερθώ σε δύο ζητήματα. Η κρίση τρέχουσα μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας, το έχουμε ξαναπεί και πάλι σήμερα είναι πρόφανες ε, πως ε, πρέπει να δημιουργήσουμε μια ανεξάρτητη αγορά ενέργειας στην Ευρώπη, ειδικά στον τομέα του αερίου, έτσι ώστε η προμήθεια αερίου και ενέργειας να μην αποτελεί αντικείμενο πολιτικών διαφωνιών. Να σας υπενθυμίσω πως η Λιθουανία πληρώνει μια τιμή 30% υψηλότερη από τους υπόλοιπους για την ε, ενέργεια. Οπότε να μιλάμε για ανταγωνισμό εντός στο εσωτερικό μιας χώρας είναι πάρα πολύ δύσκολο και έχει αυξηθεί επίσης συνολικά κατά 30%. Κατά τα λοιπά συμφωνώ πλήρως με τον κύριο Τούρμες. Πρέπει να εστιαστούμε στο ε, ζήτημα αυτό. Πρέπει να τύχει προσοχή σε αυτή την έκθεση έτσι ώστε η Κομισιόν να συστήσει μια επιτροπή που δεν ασχολείται μόνο με τις τιμές της ε, ενέργειας. Εάν συσταθεί μια τέτοια επιτροπή θα δούμε διάφορους ενδιαφέροντες ε, παράγοντες. Υπάρχουν εθνικές προτεραιότητες κάποιων κρατών μελών και πάλι στο μέλλον πρέπει να σκεφτούμε τις ανταγωνιστικές πηγές ενέργειας και να ξεκινήσουν και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα ήθελα να συμφωνήσω με την εισηγήτρια πως η σύγκρουση Ρωσίας και Λευκορωσίας πρέπει να τονιστεί πίσω κάπου στα εκτιμώντας και θα πρέπει επίσης να δώσουμε βάρος στις διασυνδέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά για να υπάρχει ασφάλεια στην προμήθεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Μπέντσαν. Δεν έχει νόημα να μιλάμε για ενεργειακή πολιτική χωρίς ε, πολιτική ασφάλειας και εξωτερική πολιτική. Όπως ε, τα βλέπω εγώ τα πράγματα, η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, από τις αγωγές αερίου θα είναι πρόβλημα, θα εξαρτώμαθε θα εξαρτώμεθα από εισαγόμενε υγιές ενέργειες από λίγε περιοχές του πλανήτη. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να βρούμε διαφορετικές πηγές και πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην ενεργειακή υποδομή σε ολόκληρη την Ευρώπη, ειδικά στη διασυνοριακή υποδομή και άρα απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις στην έρευνα και στην τεχνολογία χαμηλού άνθρακα για να είναι η Ευρώπη σε θέση να εκμεταλλευτεί καλύτερα τους ενεργειακούς της πόρους. Νομίζω πως ε, τα σχόλια που ακούστηκαν στη σημερινή συζήτηση έδειξαν πως πρέπει η ενεργειακή πολιτική να εστιαστεί περισσότερο στην αγορά και στον ανταγωνισμό. Πρέπει να φροντίσουμε πως ε, αυτό θα γίνει για να έχουμε ασφάλεια ε, ενεργειακή. Έχουμε λοιπόν προβλήματα ανταγωνισμού στην Ευρώπη, αλλά εγώ πριν από 8 χρόνια είχα διαπραγματευτεί το δεύτερο ενεργειακό πακέτο στην Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς και υπήρχαν ζητήματα με το δίκτυο και με τον ανταγωνισμό μεταξύ διαφόρων εταιριών. Πέρασαν 8 χρόνια, πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά ακόμα πρέπει να, πρέπει να γίνουν πολλά. Η ενεργειακή πολιτική επίσης πρέπει να συνεισφέρει στην ενίσχυση της ε, ασφάλειας ε, παροχής να μειωθούν ε, τα αέρια θερμοκηπίου και όπως είπε και ο κ. Στούρμες αυτό πρέπει να συνδεθεί και με την ασφάλεια της παροχής. Έχουμε λοιπόν αυτές τις δύο εκθέσεις που μιλάμε για την ενεργειακή στρατηγική σήμερα και Υπάρχει και το σχέδιο δράση για την αποτελεσματική χρήση ενέργειας και εκεί πέρα ο συγγητή λέει πω πρέπει να συντονίσουμε αυτές τις δύο εκθέσεις γιατί πράγματι αλληλεπικαλύπτονται. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την συγγήτρια να συντονιστούν αυτές οι δύο εκθέσεις. Ευχαριστώ κύριο Σκάντσεν. Θα ήθελα να μιλήσω και εγώ για αυτό το επιχείρημα για λίγο και να σας ζητήσω να βρούμε χρόνο για να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση, να δώσουμε περισσότερο χρόνο σε αυτή τη συζήτηση. Είναι ένα από τα θεμελιώδη ζητήματα της Ευρώπης για το 2020. Ε, αρνούμε να μπω στο ουσία της συζήτησης. Θα ήθελα μόνο να σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για το οποίο εσείς μιλήσατε. Μιλήσατε για τον διάδρομο 1. Ε, παρουσιάστηκε μία ολοκληρωμένη πρόταση παραγωγής, εφοδιασμού ε, και μεταφορής και μεταφοράς και διανομής, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μπορούσε να είναι ένα χαρακτηριστικό πρόγραμμα για το πώς πρέπει να αναπτύξουμε αυτή την παραγωγή και χρήση. Ε, μια ολοκληρωμένη παραγωγή και χρήση της ενέργειας. Ε, μόνο θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή ε, στη χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση πρέπει να έχει τρία χαρακτηριστικά. Ορθολογικότητα των λίγων ορθολογική χρήση των λίγων πόρων που έχουμε, χρήση των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και σωστό συντονισμό των πόρων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Χιούνα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το έγγραφο αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Νομίζω ότι όλες οι χώρες μας στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν κάποιο είδος κρίσης και θα πρέπει να προετοιμάσουμε την καλύτερη εφαρμογή της στρατηγικής για το 2020. Όπως και εδώ πέρα, δεν υπάρχουν σαφείς προτεραιότητες, έχουμε ένα μείγμα βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων πρέπει να τονίσουμε ότι είναι σημαντικό να επιλέξουμε ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί στόχοι και να τους εφαρμόσουμε στην επόμενη εννέα αιτία. Γνωρίζουμε τη σημασία του ενεργειακού προβλήματος, βλέπουμε τα προβλήματα με την τροφοδοσία σε φυσικό αέριο, βλέπουμε και τη δυνατότητα εξαγωγής φυσικού αέριου από ασβεστολιθικά σχιστολιθικά πετρώματα, αλλά οι επιστήμονες λένε ότι αυτό δεν θα είναι διαθέσιμο στο άμεσο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν για τα επόμενα χρόνια να βρούμε στόχους οι οποίοι να είναι εφαρμόσιμοι ήδη με τις σημερινές συνθήκες. Αυτό το οποίο ελείπει από την έκθεση είναι το γεγονός ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε δεν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των στόχων και από ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Οι εθνικοί προϋπολογισμοί θα, περα, θα περατωθεί η εξέτασή τους και θα οριστικοποιηθούν τον Οκτώβριο περίπου του έτους αυτού. Αν τα κράτη-μέλη δεν ξέρουν τι πόρους θα έχουν για αυτή την κατεύθυνση και δεν έχουν τη δυνατότητα να βρουν τέτοιους πόρους, θα χάσουμε το πρώτο χρόνο. Όλες οι χώρες αυτή τη στιγμή προσπαθούν να ικανοποιήσουν βραχυπρόθεσμους στόχους. Αυτό σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα δύο-τρία χρόνια θα χαθούν αν καμία χώρα δεν είναι σε θέση να εφαρμόσει αυτούς τους στόχους. Θέλω λοιπόν να τονίσω τη σημασία της επίτευξης στρατηγικών στόχων στην έκθεση αυτή. Θα πρέπει να έχουμε την κατάλληλη χρηματοδότηση η οποία θα έχει καθοριστεί ήδη το ποσοστό αυτών που θα προέλθουν από τα κράτη-μέλη και αυτών που θα προέλθουν από τον κοινωτικό προπολογισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέω ο ο κύριος Ντε έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά για την αποδοτική χρήση της ενέργειας τα επόμενα χρόνια. Η αποτελεσματική χρήση και η ασφάλεια της ενέργειας είναι δύο στρατηγικοί στόχοι για την Ευρώπη οι στόχοι της στρατηγικής για το 2020 είναι σίγουρα πολύ φιλόδοξοι. Η Ευρώπη, όπως υπενθύμησαν πολλοί, πρέπει να αποτελέσει μια ανεξάρτητη αγορά. Και η στρατηγική 2020 μας λέει ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι μας για τις εκπομπές των αερίων ε, του θερμοκηπίου, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για την, ενεργεια... για την εξοικονόμηση ενέργειας. Πρέπει να συμπληρώσουμε την εσωτερική αγορά ενέργειας και να υλοποιήσουμε ένα τεχνολογικό σχέδιο για μια ευρωπαϊκή στρατηγική της ενέργειας. Για την υλοποίηση αυτών των στόχων δεν πρέπει να χάσουμε το τρένο της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας. Παρόλο που το ενεργειακό θέμα συνάδει με πολύ ευαίσθητους γεωπολιτικούς ε, συσχετισμούς, ε, θυμόμαστε όλοι την κρίση που σημειώθηκε πριν από μερικά χρόνια. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενέργεια πρέπει να προσανατολιστεί σε τρεις στόχους. Την ασφάλεια των εφοδιασμού, τον ε, εξονυχιστικό έλεγχο των εθνικών σχεδίων και την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτός εδώ μπροστά μας είναι ένας δεκάλογος καλών προθέσεων. Δεν υπάρχει από πίσω μια σωστή στρατηγική οικονομικής στήριξης. Ε, τα διαρθρωτικά ταμεία, η πόρη συνοχής, ε, ad hoc, χρηματοοικονομικά εργαλεία λείπουν. Αυτά απαιτούνται για μια βιώσιμη, ασφαλή και ανταγωνιστική ενεργειακή πολιτική. Για την μελλοντικό οικονομικό προγραμματισμό ε, μέχρι το 2020 τι θα αλλάξει. Τι θα κάνει για τους στόχους της απασχόλησης. Θα υπάρξουν αυτά τα δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν υποτίθεται μέχρι το 2020. Θα δοθεί αυτό το 20% στην εξοικονόμηση της ενέργειας και τους ανανεώσιμου πηγές ενέργειας ο στόχος της αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας, της ασφάλειας, της απασχόλησης απαιτεί κατάλληλες οικονομικές, ε, κατάλληλες χρηματοδοτικές πολιτικές. Διαφορετικά δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Ευχαριστώ. Κύριος Ρίμπιχ, εγώ θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα τη σημασία του τομέα έρευνας και ενέργειας θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα εργαλεία τα οποία θα θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε στον τομέα της, ενέργειας, έρευνας για την ενέργεια και να βελτιώσουμε την κατάσταση στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό να δώσουμε περισσότερη έμφαση στην αποθήκευση ενέργειας, γιατί πάρα πολλές από τις τεχνολογίες τις νέες βασίζονται στη δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τις τεχνικές που έχουμε στη διάθεσή μας προς την κατεύθυνση αυτή. Η δεύτερη δυνατότητα έρευνας θα ήταν οι κοινέ πρωτοβουλίε ενέργεια σε ό,τι αφορά την ε, κατακράτηση, την ε, δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακος. Νομίζω ότι η γη δεν είναι ο καταλληλότερος χώρος για την αποθήκευση και τη συγκράτηση του διοξιδίου του άνθρακος. Επίσης θα πρέπει να δώσουμε και έμφαση στην αντιμετώπιση άλλων αερίων όπως το μεθάνιο που παράγονται από τη βιομηχανία. Ένα τρίτο σημείο είναι ότι αυτή η σκέψη για την ε, ενέργεια θα πρέπει να περιλάβει και τους τομείς χρήσης της ενέργειας. Εδώ το 8ο πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά με μια χρηματοδότηση τάξης των 50 εκατομμύριων ευρώ που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Κύριε Ούλσκοκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα σουηδικά, σουηδιστή. Είμαι σκιώδης ε, εισηγήτρια για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες και θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την παρουσίαση που έκανε στην πρώτη αυτή συζήτηση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσουμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε και φυσικά θα πρέπει να έχουμε μια μακροπρόθεσμη σχεδίαση για να μπορέσουμε να έχουμε ελπίδες ότι θα ευδοκιμήσει το εγχείρημα αυτό το οποίο έχουμε υπομειστεί. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε και νέες συγκρούσεις στον τομέα αυτό. Η ενεργειακή πολιτική είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτό το οποίο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι να βασιστούμε στους τομείς όπου υπάρχει η μεγαλύτερη συνένεση και αυτό ο αυτό συγκεκριμένο συμβαίνει στον τομέα της αύξηση τη ενεργειακή απόδοση, τη εξοικονόμηση επομένω ενέργεια. Μέχρι στιγμή όμω δεν έχουν επιτευχθεί πολλά στον τομέα αυτό. Δεν έχουν γίνει αρκετά. Γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε μια έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργεια, στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Παράλληλα όμω θα πρέπει να δώσουμε έμφαση και στι ανανεώσιμε ενέργειε. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Παραδείγματο χάρη, της επέκτασης της των ε, εναλλακτικών ενεργειών και να χρησιμοποιούνται σε εξίσου θετικές συνθήκες όσο και οι συμβατικές μορφές ενέργειας. Και εξάλλου δεν πρέπει να λησμονήσουμε τον καταναλωτή. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι υπάρχουν περιοχές στην Ευρώπη οι οποίες ζουν σε ένδια ενέργειας και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Ευρώπης αντιμετωπίζει αυτή την ενεργειακή ένδια. Δεν μπορούμε να λύσουμε σήμερα και ούτε μπορούμε, ούτε θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα στην Ευρώπη, μέσα στην Ευρώπη. Εγώ πιστεύω όμως ότι η ενεργειακή απόδοση και η μεγαλύτερη χρήση εναλλακτικών πηγών και η βελτίωση των υποδομών με τις κατάλληλες επενδύσεις είναι αυτά τα οποία είναι απαραίτητα και αυτά έχουν σημασία και από την πτυχή της πολιτικής απασχόλησης γιατί θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε την κρίση που σοβεί σήμερα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ε, η Κομισιόν να παρέμβει, κυρία Ούτμαν. Σωστά. Όχι. Χάουτμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Κομισιόν προετοιμάζει το έγγραφό της, θα είναι έτοιμο μέχρι τον Νοέμβριο. Ακούσαμε πολύ προσεκτικά την συζήτηση που ήταν νομίζω πλούσια δεν βλέπω κάτι που να απαιτεί συγκεκριμένη αντίδραση. Υπάρχουν κάποιες αποχρώσεις όσον αφορά τις ε, προτεραιότητες και θα συνεχίσουμε να σας ακούμε και να ακούμε τις αντιδράσεις στη διαβούλευση που θα τελειώσει 2 Ιουλίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Υπάρχουν ερετήσεις ε, ε, προς την εισηγήτρια πριν λάβει τον λόγο. Παρακαλώ λοιπόν, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταλλαγή αυτή των απόψεων. Είναι σαφές πως οι προσδοκίες μας ε, από την Κομισιόν διαφέρουν αρκετά γιατί ακούσαμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης κάποιες, ε, κάποιους που ζητούσαν να επανεξεταστεί το πακέτο κλίματος και ενέργειας, από την άλλη κάποιοι ζητούσαν περισσότερη έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι σαφές πως πρέπει να θέσουμε κάποιους στρατηγικούς στόχους. Η Κομισιόν το έχει ήδη κάνει αυτό, πρέπει να σκεφτούμε τους δικούς μας κοινοβουλευτικούς στόχους, όμως ε, πρέπει να είμαστε συνεπείς. Ή θέλουμε μια κοινή ενεργειακή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα εγγυάται ασφάλεια με χαμηλές τιμές ή θέλουμε να επικεντρωθούμε στην συγκεκριμένη κατάσταση του κάθε κράτους μέλους. Προφανώς ε, κάθε κράτος μέλος έχει το δικό του ενεργειακό μείγμα, όπως επισημάνθηκε, αλλά στόχο θα πρέπει να έχουμε μια κοινή αγορά ενέργειας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα επιτύχουμε χαμηλές τιμές ε, και ασφάλεια. Οπότε θα βοηθήσουμε την ε, Κομισιόν να επιτύχει τον στόχο της για να έχουμε μια κοινή πολιτική ενέργεια. Στο ζήτημα της χρηματοδότησης είναι δύσκολο, επισημάνθηκε πως ε, η στρατηγική δεν έχει κανένα νόημα εάν δεν έχει χρηματοδότηση. Πρέπει να το αναφέρουμε λοιπόν αυτό στο έγγραφο. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω πάλι όλους τους ομιλητές και αναμένω και τα γραπτά σας σχόλια τη βδομάδα που έρχεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για ε, αυτά τα οποία μας είπατε κυρία Κολονσκαποπίνσκα. Ίσως μια ακόμα παρατήρηση. Μιλήσαμε πάρα πολύ για τους στόχους εδώ πέρα και είναι εύκολο αυτό να συνεννοηθούμε για τους στόχους. Θα πρέπει ίσως να σκεφτούμε μετά πώς θα επιτευχθεί και ο κάθε στόχος, γιατί μια φορά υπάρχουν και τεχνικά προβλήματα για τα οποία πρέπει να πούμε. Μιλ, ακούσαμε σήμερα παραδείγματος χάρη πολλά για τα δίκτυα και θα μπορούσαμε ίσως ε, κάποια στιγμή να μιλήσουμε με ειδικού ή να ακούσουμε από τους ειδικού τι είναι εφικτό τεχνολογικά στα δίκτυα. Θα έχουμε πολλές προκλήσεις λόγω των ανανεώσιμων, γιατί υπάρχουν ελλείμματα ήδη σε πολλούς τομείς και η τεχνολογία δεν είναι τόσο απλή ε, για να συνδεθούν έτσι απλά τα δίκτυα. Οπότε να ακούσουμε καμιά φορά και κανένα μηχανικό και να δούμε αν είναι εφικτά αυτά τα, τα σχέδια. Θα μπορούσαμε ίσως λοιπόν να σκεφτούμε Μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε μια σύντομη φάση με τους ε, ειδικού. Βεβαίω τώρα παρεμβάλλονται οι διακοπές. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό μετά τις διακοπές. Σα ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Εδώ πέρα τελειώνει η συζήτηση. Ε, επειδή επικρατεί λοιπόν και λίγη φασαρία, κάνουμε ένα-δύο λεπτάκια διάλειμμα και θα περάσουμε στην ε, ψηφοφορία για να γίνουν και οι συζητήσεις, ε, να πάρετε τον κατάλογο των ψηφοφοριών. Λοιπόν, σε δύο λεπτά και συνεχίζουμε. Κυρίε Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα έχουμε και δουλειές. Λοιπόν, συνεχίζουμε. So, liebe... Ξεκινάμε λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι. είναι κάπως ε, εκτεταμένος ο κατάλογος, αλλά νομίζω θα τα καταφέρουμε. Ξέρετε πώς άλλαξε λίγο ο κατάλογος ε, Ξεκινάμε με την έκθεση για τα ελαφρά εμπορικά οχήματα, η έκθεση Langen δηλαδή. Αν συμφωνείτε, ξεκινάμε. Έχετε όλες τις κάρτες σας. Μία παρατήρηση μόνο ο κύριος Λάγκεν. Μία σύντομη παρατήρηση εάν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, για να εξηγήσω εδώ πέρα. Έχουμε νέα συμβαστικές ε, προτάσεις συνολικά και σε ένα σημείο υπάρχουν δύο. Αυτό αφορά τους μακροπρόθεσμους στόχους. Εγώ μελέτησα ακριβώς ποιες προτάσεις έχουν υποβληθεί και απέσυρα την ε, δική μου τροπολογία και πρότεινα ως στόχο μακροπρόθεσμο τα 150 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο. Υπάρχει και ένας άλλος στόχος, τα 140 γραμμάρια που υποβλήθηκε από δύο ομάδες. Θεωρώ πως πρέπει να λάβουμε την απόφαση εδώ πέρα με βάση όχι μόνο το τι είναι τεχνικά δυνατό, αλλά και το ποιοι είναι οι χρήστες αυτών των οχημάτων, που είναι οι μεσές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε εγώ θα πρότεινα τα 150, αλλά πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους εκ των προτέρων για τη μεγάλη ετοιμότητα που επέδειξαν για συμβασμό σόβορα. Σας ευχαριστώ. Τροπολογία 1. Κατά. Ναι, μια στιγμή, μια στιγμή, άλλη μια παρατήρηση ο κύριος Τούρμας. Ε, τώρα, για τη μεσαία τάξη εγώ το βλέπω αλλιώ, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτό το θέμα. Εξαρτάται εδώ πέρα, μετράει κάθε Ψήφο. οπότε πρέπει να μετρήσουμε νομίζω ποιοι είναι εδώ πέρα και ποιοι ψηφίζουν πριν ξεκινήσουμε. Ωραία, θα προσέχει ούτως ή άλλως η γραμματεία, αλλά μπορούμε να κάνουμε μια δοκιμή πρώτα απ' όλα, να δούμε ποιος επιτρέπεται και ποιος δεν επιτρέπεται να ψηφίσει, να περιμένουμε και την κυρία Ποδηματά και τον κύριο Βιδάλ Κουάντρας για να κάνουμε έναν έλεγχο. Ψηφίστε λοιπόν για αν είναι να διακόψουμε τη συνεδρίαση και να πάμε όλοι μαζί στην πισίνα. Ποιος είναι υπέρ. Άρχεται λοιπόν η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ναι. Ένα λεπτό και μία κάρτα λοιπόν. Έχουμε δύο από το ΕΛΚ παραπάνω. Είναι μονίμως οι ίδιοι νομίζω. Τρεις. Τρεις παραπάνω από το ΕΛΚ και η κυρία Χολ. Δεν δουλεύει το μηχάνημά μου. Μπορούμε να βοηθήσουμε την κυρία Χολ. Α, λειτουργεί. Δεν υπήρχε ηλεκτρισμός, λοιπόν. Τώρα λοιπόν είναι όλα εντάξει, οπότε παρακαλώ να ψηφίσετε. Ποιος κέρδισε? Ωραία. Λοιπόν, Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. όχι. Α, αν θέλετε, επαλήθευση. Αρκεί να μην το κάνουμε συνέχεια γιατί θα τελειώσουμε ούτε αύριο. Λοιπόν, πέρασε. Και Καλή ιδέα να το επαληθεύσουμε. Πράγματι. Απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μα δεν είπα τίποτα. Και φωνάζεται αμέσως. Δεν πρόλαβα τίποτα να πω. Ωραία ξεκινάμε. Λοιπόν, επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Όχι. Κυρία Χολ. Δεν δουλεύει πάλι το μηχάνημα. Κυρία Χόλ, τι συμβαίνει, δεν, υπάρχει ρεύμα εκεί πέρα. Ε, ήταν, πα, μου φαίνεται βασιστήκαμε σαν ανανεώσιμες. Όχι, όχι, εντάξει, με συγχωρείτε. Now? Τώρα, ούτε. Δουλεύει ή όχι. Ωραία, λοιπόν. 29 και 67 υπέρ. Κατά. Καταπίπτει, καταπίπτει, καταπίπτει. Μάλιστα. Ναι. Περνάμε στην 80 υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται παρακάτω 81 υπέρ κατά αποχές δεκτή 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 85 σε δύο κομμάτια πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές δεκτή δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 υπέρ α κατά πίπτη. δεν προσέχω 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται, εγκρίνεται. Α, να επαληθεύσουμε. Συμβαστική 2 άρχιτη ψηφοφορία λοιπόν. Κάποιος παραπάνω από το ΕΛΚ. Τώρα εντάξει. Πέρας. Ε, ναι, σαφές. Δεκτή. 87 υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 υπέρ κατά α κατά ναι έγινε δεκτή 87 οπότε καταπίπτει και όπως και 91 περνάμε στην 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνάμε στην 96, 14 επίσης, 103 άρα, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, καταπίπτει, Εκατόν τέσσερα μέχρι 107 όχι και αυτές. Λοιπόν, συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Περνάμε άρα στο μπλοκ 110 και, και εξής ως προστίκη στην συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 116 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε. Να επαληθεύσουμε. Συμβαστική 7. άρχη της Είναι ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Πέρας. Και εγκρίνεται. Ναι. 18 λοιπόν υπέρ. Κατά. Να τα ξαναδούμε σας παρακαλώ. Υπέρ του 18. Κατά. Να επαληθεύσουμε, συγγνώμη. 18 υπέρ. Πέρας. Απορρίπτεται. 122. Όχι. 50. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 129 υπέρ. Κατά. Εποχές δεκτή. 133 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 141 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 146 ναι ναι συμβαστική 4 ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία πέρας ε δίκιο είχα Ορίστε. Δεν δουλεύει. Στο νούμερο 10 πρόβλημα με το μηχάνημα. Μπορεί κάποιος να, να το δει. Υπέρ ή κατά είχατε. Νομίζω υπέρ. Τέλος δεν αλλάζει το αποτέλεσμα. 19 όχι. 150 πάει και αυτή. 166 υπέρ κατά αποχές δεκτή 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή 23 και 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 υπέρ κατά Αποχές. Δεκτή. 170 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 171 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 172 υπέρ. Κατά. Να το επαληθεύσουμε την 172 άρχη ψηφοφορία. 172. Πέρας. Απορρίπτεται. 173 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Δεκτή. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή Πολλές σελίδες παρακάτω, 28. 28 υπέρ. Α, πήγα πολύ γρήγορα. Είμαστε σελίδα 11 τη δικιά μου. 28 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 240 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 243 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 246 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Να επαληθεύσουμε ένα για τα τσίμα τσίμα. 2.46 η ηλεκτρονική σφοφορία άρχεται. Πέρας. Και όμως δεν εγκρίνεται τότε. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Να παληθεύσουμε. Συγγνώμη. 31 λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά αποχές ε, ναι, την επαληθεύσουμε οπωσδήποτε 35 άρχη ψηφοφορία πέρας δεκτή λοιπόν 2 ποιος είναι υπέρ Ε, τελείωσε τώρα. Συγγνώμη, δεν, μπορούμε να τα κάνουμε συνέχεια. Ορίστε. Εκτός μικροφώνου ένα σχόλιο. Τι, τι δεν άκουσα λέει ο πρόεδρος, με συγχωρείτε. Στην 34 ζητήσατε επαλήθευση. Μάλιστα. Ε, να, το ξανακάνουμε. Κανονικά δεν, το, δεν πάμε προς τα πίσω, αλλά επειδή δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Λοιπόν, 34 επαλήθευση. Όχι, όχι, περιμένετε. Λοιπόν, Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Και δεκτή. Ευχαριστώ. Ε, δεν δε θα τις κάνουμε όλες τώρα. Λοιπόν, δύο... Την παριθμόν δύο, ε. Δύο. Υπέρ. Υπέρ της 2 παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Να επαληθέψουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Με ισοψηφία. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρία υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή τέσσερα υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε την 4 άρχεται η ψηφοφορία πέρας και δεκτή ε, άμα δεν το κάνουμε συνέχεια τσίμα τσίμα. Λοιπόν, 44 υπέρ. Κατά. Ναι, αποχές. Απορρίπτεται. Αυτό ήταν σαφές. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό κατά εποχές δεκτή 8 υπέρ κατά εποχές δεκτό 55 μια στιγμή όχι τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική άρχεται η ψηφοφορία πέρας και είναι σαφή τα αποτελέσματα, συγχαρητήρια. Το αποτέλεσμα. Λοιπόν, με αυτό περνάμε Ποιος ε, συμφωνεί παρακαλώ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ξανά, με συγχωρείτε. Περνάμε για... Είναι μια μία και μοναδική ψηφοφορία ηλεκτρονική για αντιστάθμιση μεταξύ διαχειριστών συστημάτων κτλ. Άρχεται η ψηφοφορία, το έχουμε συζητήσει. Πέρας. Είναι ένα παραπάνω από το ΕΛΚ. Ωραία. Πέρας. Απορρίπτεται. Μάλιστα. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία για την έκθεση Μαρινέσκου. Excuse Φιγκορέδο, με συγχωρείτε. Περνάμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 1 υπέρ Υπέρ της 1. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 3 υπέρ. Κατά. Α, τσίμα τσίμα. Αποχές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται ψηφοφορία. Πέρας δεκτή 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή ε, με συγχωρείτε συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε Στη συμβαστική 1, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 14, 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά εποχές. δεκτή 11 πάει 24 συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε συμβαστική 2 άρχη τη ψηφοφορία πέρας δεκτή 28 όχι Νούμερο 12 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό καταπίπτει, καταπίπτει. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 22 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 23 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνάμε στην 29 προφορική τροπολογία. Κυρία Μαδουρέλ. Α, με συγχωρείτε. Νόμιζα πως θέλατε να πείτε κάτι. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή καταπίπτουν καταπίπτουν συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 48 υπέρ κατά αποχές δεκτή 49 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή Πέντα 54 με συγχωρείτε α ήταν έχουμε προφορική τροπολογία Ζαντό Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε στην τροπολογία αυτή <clears throat> ζητούμε να αποσυρθεί η λέξη ετικ, ηθική γιατί φαίνεται ότι δημιουργεί κάποιες παρεξήγησεις αυτή η λέξη. Καταλάβατε. Υπάρχει κάποια αντίρρηση, δεν βλέπω. Περνάμε στην ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ της 54. Κατά. Και οι λοιποί δεν έχουν όρεξη πια. <laughs> Ε, συγγνώμη, επαναλαμβάνουμε. Λοιπόν, 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α, τρίτη φορά να ψηφίσουμε αντεπαλήθευση. Για την 54 με την προφορική τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρας. Και το αποτέλεσμα είναι δεκτή. Λάθος έγινε. Κύριε Καβέλιο. Καρβάγιο. Um με συγχωρείτε τότε. Να την επαναλάβουμε γιατί δεν υπήρχε διερμηνία. Σπάνιο, αλλά... Θα ξαναπροσπαθήσουμε. Λοιπόν, με διερμηνία αυτή τη φορά. Ε, ηρεμήστε, ηρεμήστε, μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, 54 την ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά με διερμηνία. 54 λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ. Και... Πέρας. Ορίστε. Παραπάνω. Περισσότεροι από την πριν. 55 ως συμπλήρωμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ποιο δεν συμμετέχει άλλο. Λοιπόν, δεκτή. 56 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 57 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 58 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 59 υπέρ. Κατά. Να το επαληθεύσουμε. 59 υπέρ. Ε, με συγχωρείτε. Πέρας. Α, απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική. άλλη ψηφοφορία. Εντάξει. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. και πέρας. Το αποτέλεσμα είναι σαφές. Συγχαρητήρια, τέλος. Περνάμε λοιπόν τώρα. Αρκετά ψηφίσαμε για σήμερα. Ωραία, ναι. Συγχαρητήρια και τα λοιπά. Έχουμε τελειώσει και τις δύο ψηφοφορίες. Πάμε στο επόμενο σημείο. Παρακαλώ να αποχωρήσετε ηρέμως και ησύχως αυτοί που δεν θέλετε να ακούσετε τη συνέχεια. Σημείο 10. Πρόταση αλλαγή του τροπολογοποίηση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάκαμψη. Σας παρακαλώ. Κυρίε και κύριοι. Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψη. Παρακαλώ. I don't know, I didn't take, uh, die Damen und Herren, die sich noch unterhalten wollen. Όσοι θέλουν να διασκεδάσουν με άλλα μέσα, σας παρακαλώ, αποχωρήστε και αφήστε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό τον νεκρό χρόνο του επόμενου σημείου, γιατί μετά έχουμε μια επίσκεψη και πρέπει του, της, της του Υπουργού. Frau, nur Κυρία Φαν Μπρέντ, έχει το λόγο. Έχετε το λόγο. Εξηγήστε μας ποιο είναι το πρόβλημα και ποια είναι τα αποτελέσματα. Dank ehm, Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, μπροστά μας έχουμε τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ξεκινήσω λίγο με το ιστορικό. Νομίζω πως όσοι παρακολουθούν το θέμα το γνωρίζουν, αλλά είναι σημαντικό να τα ξαναπούμε πριν περάσω στην ίδια την πρόταση της ε, Κομισιόν και σας πω κάποια πράγματα για την έκθεση την οποία έδωσα χτες για μετάφραση και ελπίζω να μπορέσουμε να την συζητήσουμε πριν τις ε, διακοπές. Το ιστορικό. Το 2009 η Κομισιόν έφερε μία πρόταση για τις... Ε, όπως ξέρετε, για την οικονομική κρίση, για το τι θα γίνει με ένα κομμάτι των αδιάθετων κονδυλίων για να ενισχυθούν οι επενδύσεις σε ενεργειακά έργα. Η πρόταση της Κομισιόν κατέληξε σε τρία μεγάλα θέματα ε, σε τρεις μεγάλους τομείς επιδότησης των έργων. Πρώτα απ' όλα υποδομές φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, δεύτερον υπεράκτια αιωλική ενέργεια και τέλος η διάσημη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Εγκρίθηκε στον τριμερή διάλογο και ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, πρέπει τώρα να ε, διαθέσει τα ε, μέσα αυτά για την αποτελεσματική χρήση ενέργειας και τις ανανεώσιμες ε, πηγές. Έχουμε λοιπόν... Βλέπουμε πως είναι πάρα πολύ αποτελεσματικές αυτές οι πηγές ενέργειας, πάρα πολύ αποτελεσματικές και σε μικρή κλίμακα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την καταπολέμηση ε, της αλλαγής του κλίματος. Ε, και για τοπικέ δουλειέ που δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλη χώρα, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικέ για την οικονομική ανάκαμψη. Βεβαίως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετείχε ε, εν μέρη στην, στον τριμερή διάλογο γιατί δεν προσαρμόστηκε ανάλογα η πρόταση της Κομισιόν. Δεσμεύτηκε όμως τότε η Κομισιόν να κάνει μια δήλωση όπου θα γίνονταν δεκτό το όραμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έλεγε πως τα διάθετα κονδύλια θα πήγαιναν προς τα εκεί. Τι βλέπουμε λοιπόν σήμερα. Εκπληρώνεται αυτή η υπόσχεση, η δήλωση της ε, Κομισιόν, η δέσμευση έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. είπα αυτή την άποψη και θα το επαναλάβω αυτό. Ε, είμαστε λοιπόν εταίροι και υποστηρίζουμε την ε, Κομισιόν και σκοπεύουμε το συντομότερο δυνατό να εγκρίνουμε αυτόν τον κανονισμό και να πάμε γρήγορα στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο έτσι ώστε το όραμα αυτό να γίνει πραγματικότητα. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα αυτό το οποίο ακολουθεί είναι αποτελεσματικές προτάσεις για να χρησιμοποιηθούν αυτά τα αδιάφτα κονδύλια με τρόπο αποτελεσματικό έτσι ώστε να έχουν μεγάλο αποτέλεσμα ειδικά όσον αφορά τις ΑΠΕ και την αποτελεσματική χρήση ενέργειας όπως το Κοινοβούλιο. Η χρηματοδότηση αφορά κυρίως τοπικές και περιφερειακές αρχές με ιδιαίτερο βάρος ε, όπως λέει και η Κομισιόν ε, στις περιοχές ε, γύρω από τις πόλεις και θα είναι με την μορφή soft loans, τραπεζικών εγγυήσεων κτλ. έτσι ώστε έργα τα οποία είναι έτοιμα στις τοπικές αρχές, τους δήμους τα οποία δηλαδή μπορούν να γίνουν ε, άμεσα, να χρηματοδοτηθούν αυτά ακριβώς τα έργα. Και το μεγαλύτερο κέρδος όπως σας είπα θα είναι σε θέσεις εργασίας, ε, αυτά τα πάρα πολύ καλά έργα στις ΑΠΕ και σε πάρα πολύ μεγάλη επίδραση που θα έχουν μέσω της χρήσης αυτών των χρηματοδοτικών μέσων. Επαναλαμβάνω, συνάδελφοι, είναι πάρα πολύ καλή αυτή η πρόταση, είναι αυτό το οποίο ζητήσαμε εμείς ως κοινοβούλιο και το καθήκον μας ε, από όλες τις ομάδες και ίσως ιδιαίτερος το δικό μου γιατί βεβαίως ε, ζήτησα αυτή την έκθεση γιατί είναι ένα θέμα το οποίο αγαπώ ιδιαίτερα. Ε, πρέπει λοιπόν να εγκριθεί γρήγορα, να ολοκληρωθεί γρήγορα. και ίσως αναλόγως και με το τι θα γίνει στη Βελική Προεδρία να δοθεί μια περαιτέρω όθηση. Πρέπει λοιπόν να κινηθούμε γρήγορα. Αυτό σημαίνει πως θα βρείτε ελάχιστες τροπολογίες, κάποιες προσαρμογές δηλαδή, που δίνουν βάση στις πράσινες δουλειές Κάποιες λοιπόν προσαρμογές που θεώρησα απαραίτητες για να δώσουμε το βάση στην καινοτομία, στα καινοτόμα έργα για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και της ΑΠΕ που αποτελούν χαρακτηριστικό τμήμα της ενεργειακής μας πολιτικής για να φροντίσουμε έτσι για την καλή σύνδεση με, την υπάρχουσα, με τα υπάρχοντα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής και να έχουν ένα σημαντικό αποτέλεσμα και ζητάμε λοιπόν τα αδιάθετα κονδύλια τα οποία κάθονται θα αυξηθούν κατά 5 εκατομμύρια τα οποία θα προσθεθούν στον προϋπολογισμό. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τροπολογίες. Αναμένω τις πρωτοβουλίες των συναδέλφων. Η έκκλησή μου είναι δεν θα κουραστώ να το λέω πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιωθεί, να ενισχυθεί η πρόταση της Κομισιόν, αλλά κυρίως γρήγορα να εργαστούμε για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία στο Συμβούλιο. Και αυτό το τελευταίο δεν είναι τόσο προφανές, δεν είναι τόσο εύκολο. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη, να μην τα κατανομάσουμε, στο Συμβούλιο που θα επιθυμούσαν τα λεφτά αυτά να μην πάνε σε νέες επενδύσεις στην ενέργεια και την αποτελεσματικότητα, αλλά να πάνε στα κράτη-μέλη πίσω. Θα είναι χαζό κάτι τέτοιο και δεν θα είναι και καλό για τους στόχους ε, που έχουμε ε, στην Επιτροπή μας για την ενέργεια, την οικονομία και την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Είμαι επεμπισμένη και ελπίζω μαζί σας να μην Ε, έχουμε περαιτέρω πρόβλημα με τους προϋπολογισμούς και την κρίση, γιατί θα πρέπει να συνεχίσουμε να ε, επενδύουμε στον τομέα αυτόν. Ευχαριστώ. Ο Σας ευχαριστώ κυρία συνάδελφε. Κυρία Κάντσης, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε και την εισηγήτρια για την παρέμβασή της, με την οποία συμφωνούμε ω σκιώδης εισηγητής για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Θα ήθελα ωστόσο να δώσω ορισμένες διευκρινήσεις. Καταρχήν συμφωνώ με το χρονοδιάγραμμα, γιατί εδώ μιλούμε για ένα ενεργειακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ανάκαμψη, σε συνέχεια όσων έχουν ήδη προαποφασιστεί. Ωστόσο, τα χρονοδιογράμματα είναι όλο και πιο αυστηρά. Πρέπει λοιπόν να παρουσιάσουμε και να εγκρίνουμε προγράμματα σύντομα, αποτελεσματικά και συγκεκριμένα. Αυτό είναι μια πρώτη συνιστόσα. Καθώς διερχόμεθα και μιας πολύ έντονης κρίσης, ε, και ακριβώς σήμερα το πρωί μιλήσαμε για την ανάπτυξη της ενέργειας και της ενεργειακής πολιτικής. Όλη αυτή η συζήτηση και η κρίση ε, νομίζω ακριβώς αιτιολογούν ε, την απόφασή μας να προχωρήσουμε Προ τι αναλλακτικέ πηγές ενέργειας, την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας κτλ. Πέρα από το χρονοδιάγραμμα υπάρχει στρατηγική ουσία. Μιλάμε για αποτελεσματική χρήση της ενέργειας, ιδίως στις αστικέ περιοχές. Αυτό είναι δεδομένη της σημασία ε, του θέματος, το οποίο εναρμονίζεται με την οδηγία ε, που εκδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα για την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας στην, στις οικίες. Επιτρέψτε μου να, να μιλήσω για τη διάσταση των προγραμμάτων, για το μέγεθος των προγραμμάτων, ε, να μειώσουμε λίγο το ποσοστό για να αναπτύξουμε περισσότερα προγράμματα. Το ποσό που έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι πολύ μεγάλο. Καλό θα ήταν λοιπόν να προσπαθήσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό προγραμμάτων, μειώνοντας τη χρηματοδότηση στο 50% και φυσικά λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική ισορροπία που είναι πάντα σημαντική. Ασφαλώς θα προσπαθήσουμε να μην επιστρέψουν οι πόροι αυτοί στα ταμεία των κρατών μελών, γιατί αυτό θα ήταν ένα βήμα προς τα πίσω. Όσο αφορά τώρα τα εργαλεία. Έχουμε τους χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Νομίζω ότι εδώ χάσαμε μια πολύ καλή ευκαιρία στο πρώτο τμήμα, στο προηγούμενο κανονισμό. Θα έπρεπε να έχουμε οικοδομήσει ένα ειδικό ταμείο ένα ταμείο που θα αποτελούνταν από, χρηματι... από οικονομικές ε, πρωτοβουλίες για τον πολλαπλασιασμό των λίγων πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να προβούμε σε ένα άλμα ποιότητας ε, σε συγκεκριμένα σχέδια. Εδώ πιστεύω ότι με αυτό το εναπομείνον ποσό που έχουμε, δυστυχώς ε, ε, αυτή η οδός έχει κλείσει μάλλον. Επομένως, ε, πλέον μιλάμε για εργαλεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία μας προτείνονται εδώ, και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επανεκκινήσουμε, να ξαναθέσουμε σε κίνηση την ενεργειακή οικονομία προς τις κατευθύνσεις τις οποίες έχουμε προτείνει. Συμφωνώ απόλυτα με όλα όσα υπόθηκαν και είμαστε στη διάθεσή σας για να συμβάλλουμε και να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα. Γιατί αυτό είναι και ο κύριος στόχος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω... Α, ο κύριος Τούρμες θέλει να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία εισηγήτρια. Νομίζω ότι αυτό που επήγε περισσότερο ε, στο θέμα αυτό είναι να ψηφίσουμε γρήγορα στην Επιτροπή μας για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Η πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω είναι πολύ καλή. Δεν βλέπω, και, δεν βλέπω μεγάλη ανάγκη για τροπολογίες. Και η ιδέα που βρίσκεται από πίσω. Ε, εντάξει, έχουμε μόνο 150 εκατομμύρια ή πάνω κάτω τόσο. Αν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε ένα χρηματοοικονομικό μέσο που να δημιουργήσει μόχλευση, ε, νομίζω ότι θα είναι καλό. Ε, είχα συναντήσεις ε, με το KFW και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που είναι δύο από τις τράπεζες οι οποίες θα διαχειριστούν αυτό το, αυτούς τους πόρους. Μου εξήγησαν οι εκπρόσωποι των τραπεζών αυτών ότι έχουν πείρα με αντίστοιχους πόρους για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βασικά είχαν πάρει χρήματα από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό Ε, είχαν αναλάβει εκείνο το κομμάτι που ενείχε τον μεγαλύτερο κίνδυνο και στη συνέχεια απευθύνθηκαν σε άλλες τράπεζες και ακριβώς σύμφωνα με αυτό που προτείνατε με τις, μέσω των συμπράξεων ιδιωτικού και δημοσίου γιατί έτσι καλύπτεται και λιγότερος κίνδυνος σχημάτισαν ένα πακέτο που ήταν λιγότερο επικίνδυνο. Τώρα, εν ώψη και αυτής της χρηματοοικονομικής κρίσης που διανύουμε, ε, πρέπει να υπερβληθούν τα εμπόδια έτσι ώστε να ε, πάνε οι πόροι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανησυχούν πάρα πολύ για τα λειτουργικά τους έξοδα. Και βασικά αποφάσισαν τα ιδρύματα αυτά να μην μειώσουν το ύψος των δανείων. Ωστόσο, αναλύουν προσεκτικά την κατάσταση και τους κινδύνους και εάν το ταμείο αυτό, εάν οι πόροι αυτοί αναλάβουν τμήμα του κινδύνου, τότε οι τοπικές τράπεζες πιο εύκολα θα μπορέσουν να συμμετέχουν και αυτές και να χορηγήσουν χρήματα για τα σημαντικά αυτά έργα για την ανακαίνιση των κτηρίων, για τους έξυπνους μετρητές, για πιο αποδοτικές συσκευές κτλ. Αυτή είναι λοιπόν η ιδέα, να δημιουργήσει κανείς ένα οικονομικό εργαλείο το οποίο να μοχλεύσει πόρους στην αγορά έτσι ώστε η πρόσβαση στο κεφάλαιο για τους επενδυτές που θέλουν να ασχοληθούν με την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας να είναι πιο εύκολο είναι πιο εύκολη. Νομίζω ότι είναι μια καλή πρόταση και πρέπει να προσπαθήσουμε να την επιταχύνουμε. Για τις εθνικές κυβερνήσεις τώρα, όλοι μας έχουμε επαφές με τις εθνικές μας κυβερνήσεις. Νομίζω ότι έχουμε μια καλή κατάσταση μπροστά μας. Αν μια εθνική κυβέρνηση θέλει να κάνει κάτι παρόμοιο, θα τις κόστιζε. Αν και τα 27 κράτη-μέλη θα έπρεπε να συστήσουν εθνικά ταμεία για να δώσουν όθηση σε τέτοιες επενδύσεις. Αυτό θα ήταν πιο δαπανηρό από τη δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού Ταμείου που θα χρησιμοποιούσε αυτούς τους πόρους του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Νομίζω για τη Βρετανία, για τη Γαλλία, για τη Γερμανία ισχύει. Αυτό για όλους τους, ε, για τους προϋπολογισμούς όλων των κράτων μελών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Φωνής Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα αυτό το οποίο έχουμε ενώπιόν μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να μπορέσει μέσω αυτού του πλαισίου να δημιουργήσει σχέδια σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα οποία έχουν θετικό αντίκτυπο σε, στην ευρωπαϊκή οικονομία στο μέλλον. Εμείς υποστηρίξαμε ιδιαίτερα το τμήμα αυτό της ενεργειακής αποδοτικότητας, το οποίο τονίστηκε και από την εισηγήτρια. Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν ένα χαρακτήρα καινοτομία. Είναι καινοτόμο και ο τρόπο με τον οποίο τίθενται στη διάθεση τα χρήματα, οι επενδύσει, ιδίω σε καιρό οικονομική κρίση. Τη στιγμή που βλέπουμε ότι οι τράπεζες διστάζουν να δώσουν κονδύλια στην αγορά, αυτό είναι ένας πολύ καλός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες της αγοράς. Μπορούμε λοιπόν έτσι να προωθήσουμε την ε, καινοτομία στον τομέα αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό, ιδίω με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και είναι μια αξιέπαινη πρωτοβουλία και φυσικά νομίζω ότι το κείμενο θα πρέπει να αναφέρει και τη δυνατότητα θετικής συνέργειας και με τα άλλα διαρθρωτικά ταμεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια ευρεία προσέγγιση γιατί έχουμε και την ε, πρωτοβουλία των Δήμων και Κοινοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα ζητήματα αυτά. Ήταν μια δήλωση η οποία νομίζω ότι είχε μια ευρεία βάση <clears throat> και έχει σαν στόχο να επιτύχουμε τους στόχους μας για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος ακόμα και πριν από το 2050. Αυτοί λοιπόν που έχουν υπογράψει αυτή τη συμφωνία μεταξύ Δήμων και Κοινοτήτων μπορούν τώρα να τύχουν χρηματοδότησης και μετά από όλα αυτά που έχουμε πει για το, την πρωτοβουλία του 2020 νομίζω ότι μπορούν να συνδυαστούν με αυτή την πρωτοβουλία και έτσι δεν έχουμε μονάχα την παρουσία των κρατών μελών αλλά και τις περιφέρειες της Ευρώπης, τους δήμους, κοινότητες, αστικές περιοχές, μια αποκεντρωμένη μορφή εταιρικών σχέσεων και αυτό είναι ένας περαιτέρω στόχος που θα πρέπει να υπάρχει στην πορεία μέχρι το 2020. Αυτό το κομμάτι ήταν κάτι το οποίο έλειπε στη στρατηγική της Λισαβόνας, η οποία στρατηγική Λισαβόνας φαινόταν ότι ήταν απλώς μια υπόθεση των κρατών μερών. Αν δεν προχωρήσουμε όμως σε επίπεδο πόλων και τοπικών αρχών, και δεν έχουμε την υποστήριξη των τοπικών φορέων, δεν θα έχουμε πραγματική πρόσβαση στους πολίτες και θα τους κινητοποιήσουμε για να προχωρήσουν στο δρόμο της καινοτομίας. και έτσι οι πρωτοβουλίε τη Κομισιόν, οι πρωτοβουλίε Ναυαρχίδο, ούτω ή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσουν να ευδοκιμήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τίκαου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι όπως και ο κύριος Φανίστλεροι θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία που επέχουν οι επενδύσεις για να έχουμε μια μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση στα κτίρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι αυτοί λοιπόν οι δρόμοι για την βελτίωση της ε, επενδύσης των, ε, της αποδοτικότητας μπορεί να είναι θετική. Τα 150 αυτά εκατομμύρια λοιπόν μπορούν να επενδυθούν γρήγορα σε στόχους ενεργειακής απόδοσης, καλύτερης μόνο στα σπίτια κτλ το Μάρτιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε ήδη αναγνωρίσει σαν στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το να υπάρξει μια βελτίωση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης μέχρι το 2020. Ξανατόνισε το Συμβούλιο ε, τον στόχο αυτό στη συνεδρίασή του του Ιουνίου. Επομένως θα πρέπει να περιμένουμε τώρα από την Κομισιό να υποβάλει συγκεκριμένε προτάσεις ώστε να μπορέσει να ανέλθει η ενεργειακή απόδοση κατά 20% μέχρι το 20, Νομίζω ότι η πρωτοβουλία ξύπνιας πόλης μπορεί να συνεργαστεί με την πρωτοβουλία αυτή προς την κατεύθυνση αυτή. Θέλω επίσης να τονίσω ότι δεν πρέπει αυτό να είναι μια απομεμονωμένη πρωτοβουλία. <clears throat> Αν θυμόμαστε, τον Απρίλιο του 2009 είχαμε τροποποιήσει τον κανονισμό που αφορούσε την περιφερειακή ανάπτυξη με στόχο να επιτρέψουμε σε όλα τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν ένα τμήμα 4% συγκεκριμένα του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για να εξασφαλίσουν την ενεργειακή απόδοση των καταλημάτων, των κτίριων λοιπόν, αλλά στα οποία περιλαμβάνονται πάντα και οι, τα κοινωνικά καταλήμματα τα οποία δημιουργούν τα κράτη-μέλη. Ακόμα όμως δεν, έχουμε, δεν έχει εγγραφεί αυτό στον προϋπολογισμό, μέσα στα πλαίσια λοιπόν τη ε, μεταρρύθμιση του προπολογισμού θα πρέπει η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν την ευκαιρία για να <clears throat> χρησιμοποιηθεί αυτό το 4% του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ακριβώς για το στόχο της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτίριων, ιδίως των καταλήμματων. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν έχει τώρα το λόγο. Κύριο Μπερούτσι, αν συμφωνείτε, μια σύντομη παρατήρηση από την Κομισιόν, αν θέλετε να κάνετε. Στο σημείο αυτό κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω απλώς να ευχαριστήσω τους κοινοβουλευτικούς για την υποστήριξη που έχουν δώσει στην Κομισιόν. Για μας είναι κεφαλαιόδηση η χρόνηση των προσπαθειών, όπως τονίστηκε και από την εισηγήτρια. Ο πολλαπλασιαστικός αυτός ρόλος που αναφέρθηκε επίσης θα είναι σημαντικός αν μπορέσουν τα μη εκταμιευμένα κονδύλια αυτού του ταμείου να συμπληρωθούν με κονδύλια από άλλες πηγές, αυτό θα οδηγήσει σε μια κρίσιμη μάζα η οποία θα είναι μικρή μεν, αλλά σημαντική, θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε σε πειράματα αυτού του είδους και θα έχουμε και αντικτύπους οι οποίοι δεν θα είναι μεμονωμένοι, όπως δεν πρέπει να είναι μεμονωμένες οι πρωτοβουλίες μας. <clears throat> έχουμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν την επόμενη ε, σειρά δημοσιονομικών προοπτικών όπου μια τέτοια επιτυχία σε αυτά τα εγχειρήματα θα έχει επιπτώσεις θετικές. Πρέπει λοιπόν να λειτουργήσουμε όλοι για να μπορέσουν τα εγχειρήματα αυτά να στεφθούν γρήγορα από επιτυχία και αυτό απαιτεί και μια λήψη απόφαση μέχρι το τέλος του ενεστώτος έτους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Φαν αν θέλετε να λάβετε και πάλι το λόγο. Εν συντομία, τις επόμενες εβδομάδες θα έρθω σε άτυπες επαφές με διάφορα μέλη της ομάδας για να καταλήξουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε κάποια απόφαση για αυτό το θέμα. Και εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο Ευχαριστώ όλους που έλαβαν μέρος σε αυτή την συζήτηση. Τον Ιούλιο θα επανέλθουμε στη συζήτηση επί της εκθέσεως της κυρίας Φανμπρέμπτ. Έχει κλείσει και αυτό το σημείο. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η συνάντηση με την Ισπανίδα Υπουργό, η οποία θα εκπροσωπηθεί από τον Υφυπουργό της, ο οποίος όμως και αυτός δεν έχει φτάσει. Έχουμε λοιπόν ένα προβληματάκι. Μπορείτε να δείτε αν είναι πρώτον πυλών ο Ισπανός Υφυπουργός, παρακαλώ. Καμιά φορά δεν θέλουν να μας ενοχλήσουν οι καλεσμένοι μας και περιμένουν υπομονετικά στην πόρτα.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 πρέπει να κάνουμε μια σύντομη διακοπή. Δεν ξέρω πότε θα έρθει όμως ο Ισπανός Υπουργός. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Η Ισπανική Προεδρία έρχεται από το αεροδρόμιο, αλλά ενδιαμέσως καταφέραμε ο κύριος ε, Βιδάλ Κουάδρας ως guest star ουσιαστικά να είναι πιο νωρίς για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το σημείο της ημερήσιας διάταξης το δικό του το οποίο είναι, έχει, θα προταχθεί με αυτόν τον τρόπο. Θέλουμε να του δώσουμε λοιπόν ένα αριστείο ταχύτητο σε ό,τι αφορά την προσέλευσή του και γι' αυτό θα δώσω το λόγο στον κύριο Βιδαλ Κουάδρας για να μας αναφέρει πώς ε, βαίνουν τα πράγματα με την οδηγία σε ό,τι αφορά τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο. Έχετε το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μου είπανε <clears throat> ότι στις 12 θα έρχονταν το σημείο αυτό της ημερησίας διάταξης. Έτρεξα όμως, σπριντάρισα όσο μπορούσα πιο γρήγορα από το γραφείο για να έρθω εδώ. Ευχαριστώ. Θέλω να ξεκινήσω ευχαριστών εκ βάθους καρδίας όλους τους κοιόδης εισηγητές και εσάς, κύριε Πρόεδρε, για την συνεχή προσφορά ιδεών και συστάσεων τους τελευταίους δέκα μήνες, από τη στιγμή δηλαδή που ξεκινήσαμε την νομοθετική διαδικασία σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για, την, για τον εφοδιασμό σε φυσικό αέριο. Πιστεύω ότι αυτό ακριβώς χρειαζόταν ένα είδος στενής συνεργασίας που έχει συμβάλει πάρα πολύ σε αυτό το οποίο ταπεινοφρόνος μπορώ να πω ότι είναι ένα επιτυχές αποτέλεσμα. Τη Δετάρτη το βράδυ φτάσαμε σε μια άτυπη συμφωνία με το Συμβούλιο στον τριγωνικό διάλογο σε σχέση με τον κανονισμό αυτό. Το κείμενο της συμφωνίας θα διανεμηθεί σε όλους σας σήμερα μόλις πάρουμε το πράσινο φως από την υπηρεσία νομικών μεταφραστών. Το Συμβούλιο θα εγκρίνει, αναμένεται μάλλον να εγκρίνει αύριο στο επίπεδο της Κορεπέρ το κείμενο αυτό και εμείς στην Επιτροπή μας ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να υπερψηφίσουμε αυτό το κείμενο τον Ιούλιο, στην επόμενη μας συνεδρίαση. Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια καταρχήν θα λάβει χώρα την δεύτερη σύνοδο Ολομέλειας του Σεπτεμβρίου. Θέλω να ευχαριστήσω περαιτέρω και την Κομισιόν για τη θαυμάσια εργασία της, ιδίω στη διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο νομοθετικών σωμάτων και θέλω να ευχαριστήσω και την Ισπανική Προεδρία για το γεγονός ότι σε πραγματικό χρόνο μας κρατούσε πάντα ενήμερους σε σχέση με την πρόοδο που είχε επιτελεστεί στους κόλπους του Συμβουλίου. Είναι χρήσιμο λοιπόν πάρα πολύ να έχουμε αυτές τις διαρροές πληροφοριών από τη συνεδριάση του Συμβουλίου. Αλλά αυτό δεν ήταν αποτέλεσμα κατασκοπίας, ήταν θεμητές παροχές πληροφοριών από πλευρά της Κομισιόν. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε πολύ καλά ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα αυτών των διαπραγματεύσεων και από τη στιγμή που θα εφαρμοστούν αυτές οι διατάξεις νομίζω ότι θα μειώσουν σημαντικά το ευάλωτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περαιτέρω διαταραχές της παροχής φυσικού αερίου με την εφαρμογή του προτύπου νη 1, με την εισαγωγή τεχνολογιών ανάδρομης ροής σε όλους τους διασυνδετές μεταξύ κρατών μελών στα επόμενα τρία χρόνια. Θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτό. Και θέλω επίσης να τονίσω και τον ενισχυμένο ρόλο της Κομισιόν για το συντονισμό δράσεων εκτάκτου ανάγκης και την ύπαρξη μιας ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο και επίσης περαιτέρω τη δυνατότητα της Κομισιόν να εξασφαλίσει ότι τα εθνικά προληπτικά σχέδια δράσης δεν θέτουν εν αμφιβόλο την ασφάλεια εφοδιασμού άλλων κρατών μελών. Γιατί αυτό ήταν ένα από τα κέρια σημεία της συζήτησης. Ότι η Κομισιόν έχει τις εξουσίες για να μπορέσει να παρέμβει σε αυτά τα προληπτικά σχέδια δράση των κρατών μελών για να διασφαλίσει την ασφάλεια φοδιασμού για όλα τα κράτη-μέλη. Και φυσικά το πνεύμα αυτό αλληλεγγύης, το οποίο είναι απαραίτητο να πριτανεύει, ώστε <clears throat> όταν έχουμε κάποια κρίση, τα κράτη-μέλη και ιδίως αυτά τα οποία επηρεάζονται περισσότερο από την κρίση, θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε επαρκείς ποσότητες φυσικού αερίου για τους καταναλωτές που χρειάζονται οπωσδήποτε να έχουν εφοδιασμό. Έχουμε εισαγάγει μια σειρά απορρίτρες σε ό,τι αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού που υπογραμμίζουν την βασική σημασία της δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία πρέπει να αναλάβει δράση για να, απο... να εμποδίσει ε, άνοδο των τιμών όταν υπάρχει στενότης τροφοδεωσίας. Να μην λοιπόν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στα κρατημένη λόγω αυτών των κρίσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα. Γιατί βλέπουμε και πάλι να αναδύεται μια νέα κρίση μεταξύ της Ρωσίας και της Λευκορωσίας. Αν αυτή η κρίση δεν επιληθεί λοιπόν, θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρό αντίκτυπο στα βαλτικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδεχομένω και στην Πολωνία. Ευτυχώς η Κομισιόν έχει ήδη αναλάβει δράση με μεγάλη ταχύτητα. Χθες ο Γενικός Διευθυντής Ενέργειας πέταξε στο Μίνσκ και ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσει να επιληθεί αυτή η κρίση το ταχύτερο δυνατό. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι διότι επιτύχαμε σημαντικές συμβιβαστικές λύσεις σε σχέση με την ενσωμάτωση των λεγόμενων νησίδων φυσικού αερίου στο δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν ρήτρε για προορισμό και αυξανόμενη διαφάνεια σε ό,τι αφορά την παροχή φυσικού αερίου στα κράτη-μέλη και μόνο με τέτοιες πληροφορίες, με γενική παροχή πληροφοριών μπορούν να λυθούν τα προβλήματα αυτά και να λυθούν οι καλύτερες απαντήσεις. Από την πλευρά του Κοινοβουλίου επίσης υπογραμμίζεται ότι η καλύτερη, τα καλύτερα προστατευτικά τείχη, οι καλύτερες γραμμές άμυνας είναι οι αγορέ. Και αυτό τώρα αντανακλάται στο κείμενο της Κομισιόν. Υπήρξε ένα σημείο το οποίο ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητο για πολλούς από του συναδέλφου μα, Το ότι η Κομισιόν έχει τη δυνατότητα να κηρύξει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κατάσταση ανάγκη και αυτό μπορεί να γίνει με πολύ μεγάλη ευελιξία. Δηλαδή υπάρχουν έχουν αρθεί τα κατόφλια τα οποία είχαν θεσπιστεί προηγουμένως και η Κομισιόν μπορεί να χρησιμοποιήσει και να ενεργοποιήσει όλους τους μηχανισμούς που προβλέπονται ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Μπορεί να πρόκειται για ένα κράτος μέλος, μπορεί να πρόκειται για πολλά κράτη-μέλη ή μπορεί να είναι περιοχές οι οποίες συνδέουν διάφορα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει ένας πάγιος ορισμός λοιπόν, επομένως η Κομισιόν έχει ένα ευρύ περιθώριο εκτίμησης βάσει του οποίου μπορεί να δράσει. Ο κανονισμός αυτός λοιπόν είναι μια πραγματική λύση σε ένα ουσιαστικό πρόβλημα. Θα προωθήσει την ε, κατασκευή υποδομών σε, τοπικό, σε εθνικό επίπεδο, τις διασυνδέσεις επίση μεταξύ των κρατών μελών και θα θεσπίσει ελάχιστα πρότυπα τροφοδοσίας για όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Τέλος, θα επιτρέψει την ταχεία, τον ταχύ συντονισμό των απαντήσεων σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης και έναντι τρίτων χωρών. Και σε σχέση με την αρχική θέση που είχε πάρει το Συμβούλιο, που ήθελε απλώς να εκδοθεί μια οδηγία στον τομέα αυτό και όχι ένας κανονισμός, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε διατρέξει μακρό δρόμο, έχουμε ένα ισχυρό κανονισμό, ο οποίος είναι και τεχνικά εμπεριστατωμένος. Και επομένως η συστασή μου αγαπητοί συνάδελφοι είναι προφανώς να υπάρξει από σας πλήρης υποστήριξη της συμβαστικής αυτής λύσης όταν ψηφίσουμε τον Ιούλιο και πιστεύω ότι από τη στιγμή που θα διαβάσετε το κείμενο που έχει την υποστήριξη όλων των σχεδόν εισηγητών θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι θα πρέπει να υπερψηφιστεί αυτό το κείμενο. Βέβαια είμαι στην απόλυτη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις, εάν το επιθυμείτε, από τη στιγμή που θα έχετε διαβάσει το κείμενο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βίλα Βιδάλ Κουάδρας για την πρώτη σας αυτή παρουσίαση και για την εξαιρετική εργασία που φέρατε σε πέρας. Ήταν δύσκολη εργασία. Μπορεί να ήταν και κουραστική σε κάποιο βαθμό και ανιαρή, αλλά σίγουρα έχει αποδώσει κάποιους καρπούς. Ο κύριος Μετσάρος έχει καταρχήν το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τη δουλειά του κυρίου Βιδαλκουάδρας και του οφείλουμε ευχαριστίες ε, για τις ε, προσπάθειές του. Προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε και όσο μπορούμε. Για τις χώρες Κεντρικής Ευρώπης είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και καλωσορίζουμε τις ε, περιφερειακές δομές περιέχοντες στο παράρτημα 4. Μας ενθαρρύνουν ενθαρρύνουν τις χώρες ε, στις οποίες ε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία διασύνδεση. Εξακολουθούμε να είμαστε όλο και πιο εκτεθειμένοι στις αγορές ε, του αερίου καθώς η ζήτηση αυξάνεται και θα χειροτερεύουν τα πράγματα εάν συνεχίσει να κόβει την παροχή η Ρωσία, οπότε δεν μπορούμε να βασιστούμε σε κάποιες ε, ικανοποιητικές λύσεις ε, και νομικές λύσεις ε, με την τρευσοδηγία. Οπότε η εσωτερική αγορά θα παίξει έναν κεντρικό ρόλο. Οι εταιρείε παροχής αερίου θα μπορούν να απευθυνθούν στους ε, πολίτες της ε, Ένωσης, στους καταναλωτές και βεβαίως χρειάζονται ανταγωνιστικές εθνικές αγορές για να μην έχουμε στρεβλώσεις και να βασιζόμαστε σε διάφορες πηγές και διαδρομές και αυτή η πρόταση είναι αναγκαία γιατί αν μια χώρα υπογράψει μια μονομερή συμφωνία μπορεί να διακινδυνεύσει η παροχή αερίου στην Ένωση. Επίσης οι χώρες θα πρέπει να βρουν πιθανές ε, ελλείψεις ε, στην ε, παροχή αερίου τις οποίες θα πρέπει να καλύψουν σε περίοδους κρίσης. Η ασφάλεια λοιπόν παροχής θα απαιτήσει μέτρα όπως η αλλαγή καυσίμων γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μειώσουμε τη ζήτηση αερίου πρέπει να συντονίσουμε τις ε, δράσεις μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν θέλουμε να αποφύγουμε ένα κενό που θα δημιουργήσει κρίση. Υπάρχουν κάποιοι τομείς ε, στους οποίους θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε το φυσικό αέριο πηγή στην ε, παραγωγή ηλεκτρισμού και έτσι να μειωθεί η ζήτηση. Ευχαριστώ. Κλοντ Τούρμες. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον Αλέχο. Λίγοι. Αυτό το οποίο λίγοι ξέρουν είναι πως το πρόβλημά μας πριν τις τελευταίες διαπραγματεύσεις την Τρίτη ήταν πως οι κυβερνήσεις δεν ήθελαν η Κομισιόν να παίξει ρόλο να εποπτεύει τα εθνικά σχέδια ανάγκης και κινδυνεύαμε να καταλέξουμε με πλημελή ευρωπαϊκό συντονισμό. Και ήταν δύσκολο να δούμε πώς θα μπορούσαν να μετακινηθούν οι κυβερνήσεις. Και μετά ο Αλέχο είχε την έξυπνη ιδέα να χρησιμοποιήσει τις διασυνδέσεις του στη Ρωσία έτσι ώστε να τύχει το θέμα περισσότερης πολιτικής ε, προσοχής πριν από τις διαπραγματεύσεις Τρίτης. I ε, Και νομίζω πως ε, λειτουργήσαν τα πράγματα και άρα από χτες το βράδυ η Gazprom ξαναγέμισε εκεί τους αγωγούς. Μπράβο, μπράβο. <laughs> Ja, das war mir auch Ich danke für den Hinweis. Das hatte ich nicht mitbekommen. Ναι, και εγώ δεν το είχα μάθει αυτό. Ευχαριστώ που μου το είπατε πως είχαμε τόσο έξυπνες ιδέες για να καταλήξουμε σε κάποια αποτελέσματα, αλλά έτσι εξηγούνται όλα. Λοιπόν, φανίστε Ρόι. Κύριε Πρόεδρε, μετά από αυτήν την τελευταία συνεισφορά, ε, δεν, ξέρω, κάποια στιγμή πρέπει να, να τελειώσουν ε, ίσως οι, οι υπερβολές, γιατί βεβαίω είδαμε και την έξυπνη πρόταση, είδαμε τα αθλητικά κατορθώματά του σήμερα το πρωί. Θέλω να σοβαρευτούμε λίγο. Πλέον δεν μιλάμε για το υπόβαθρο, μιλάμε για το αποτέλεσμα και το δείχνει αυτό η επικαιρότητα αυτή τη εβδομάδα. καθώς χρειαζόμαστε μέσα για να αποκτήσει και μια πρακτική μορφή αυτή η αλληλεγγύη και υπάρχει τώρα η ομάδα συντονισμού αερίου που παίζει σημαντικότερο ρόλο και υπάρχει μια σαφής περιφερειακή διάσταση για όσον αφορά την αγορά αερίου και με αυτή την πρόταση συμπληρώνουμε αυτό το οποίο είχε ζητήσει ο Μπουζέκ, δηλαδή να κινηθούμε σε Ευρωπαϊκή Ένωση, να κάνουμε κάποια βήματα σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό κάνουμε λοιπόν Δίνουμε λοιπόν ένα περιεχόμενο στην αλληλεγγύη, στι διασυνδέσεις και στη συνεννόηση μεταξύ μας, πράγματα τα οποία πρέπει πράγματι να γίνουν και ακριβώς αυτές ε, οι προτάσεις δείχνουν πως ε, χωρίς να γίνονται όλα με κεντρικό τρόπο μπορούμε να συνεργαστούμε και όταν έχουμε μια κρίση. Μέσω μιας τέτοιας κρίσης μπορούμε να αλλάξουμε τρόπο σκέψης, ε, για την αποτελεσματικότητα του συστήματος παροχής ε, αερίου. Πράγματι είναι, είναι κάτι το σημαντικό αυτό που παρατηρούμε. Είναι η διασύνδεση του δικτύου φυσικού αερίου μια σημαντική υπόθεση. Οπότε συμφωνώ και εγώ με το αίσθημα του κυρίου Τούρμες. Ο κύριος Φιντάλ Κάντρας πραγματικά ήταν ε, σε αυτό συμφωνούμε όλοι, εξαιρετικός. Μια που είμαστε στις ευχαριστίες, να ευχαριστήσω και τους διαφορούς συνεργάτες εδώ πέρα που εργάστηκαν στη γραμματεία, στους βουλευτές, το Συμβούλιο και την Κομισιόν οπωσδήποτε πρέπει να ευχαριστήσουμε γιατί την ξεχνάμε συνεχώς. Μεταξύ των διαφόρων ημερών και ωρών που περνούσαν πάρα πολλοί βοηθοί και συνεργάτες ε, διαπραγματεύτηκαν και μας βοήθησαν και πρέπει να τα πούμε αυτά. Ο κύριος Σιμάνσκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Έκανε πραγματικά πολλή δουλειά, μεγάλη προσπάθεια. Ο κανονισμός αυτός έχει μεγάλη σημασία Προφανώς στόχος μας είναι ένας συμβιβασμός ο οποίος θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε προσδοκίες που ήταν διαφορετικές και πιο φιλόδοξες ήταν κάπως πιο φιλόδοξο το κοινοβούλιο και εδώ πέρα διαφωνούσε π.χ. το Συμβούλιο στην αντιστροφή της ροής, παραδείγματος χάρη. Ήταν ε, κάποιες διατάξεις, οποίες επέμενε το Συμβούλιο ότι θα σημαίνουν ε, ότι υπήρχε σε έναν συγκεκριμένο αγωγό δεν ήταν δυνατή η αντιστροφή της ε, ροής λόγω πολιτικής πίεσης από τη Ρωσία. Ένας αγωγός ο οποίος θα κλείσει αν δεν πάνε καλά τα πράγματα. Εμείς προτείναμε λοιπόν κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο. Μιλάω για τις ρήτρες επανεξαγωγής και τις ρήτρες προορισμού. Αλλά καταλήξαμε τελικά σε κάτι πολύ γενικότερο. Ας ελπίσουμε πως δεν θα οδηγήσει σε μια κατάσταση στην οποία η Κομισιόν θα αισθανθεί τώρα πως δεν έχει πλέον καθήκον να ταχθεί κατά ε, των λύσεων της αγοράς. Επίσης έχει σαχθεί μετά από τις διαπραγματεύσει και η περιφερειακή διαχείριση κρίσεων, αλλά θα πρέπει να διασφαλίσουμε πως δεν θα δικηθούμε έτσι σε μια κατάσταση στην οποία ε, δεν θεωρεί αυτόν ε, υπεύθυνο η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις περιφερειακές κρίσεις. Εξάλλου επηρεάζεται ολόκληρη η περιφερειακή κρίση από οποιαδήποτε διαταραχή της παροχής αερίου. Εξάλλου έχουμε νομικά μέσα τα οποία δεν ε, σημαίνει οπωσδήποτε πως υπαρχούν, και νομική εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ πέρα έχει εξασθενήσει αυτή από το Συμβούλιο και το Συμβούλιο έχει κάνει λάθος ε, το να περιορίζει συμμετοχή μας σε πολιτικά ζητήματα και ζητήματα εξωτερικών σχέσεων. Ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει, πως θα αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε μελλοντική κρίση αερίου ως ένα καθαρά εμπορικό ζήτημα. Αυτά τα ζητήματα έχουν και πολιτική διάσταση. Και μια κυβέρνηση, συνήθως μια κυβέρνηση στα ανατολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αντιμετωπίσει πολιτική δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώ, θα φανούμε αδύναμοι. Σε γενικέ γραμμέ όμως είναι καλή η συμβαστική λύση. Καταφέραμε να διατηρήσουμε αρκετές ε, θετικές διατάξεις. Κυρία Ρέιρα Μαδρουέλη. Ευχαριστώ πολύ κυρία, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Σφόμποντα, ο εκπρόσωπος ομάδας μας, είναι στο κτίριο αλλά δεν μπόρεσε να έρθει πιο νωρίς γιατί προβλεπόταν να γίνει αυτή η συζήτηση στις 12. Είναι όμως μια ευκαιρία για μένα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον κύριο Βιδάλ Κουάδρος για το έργο του και επίσης και να τον ευχαριστήσω για τα πολύ θετικά του λόγια για την Ισπανική Προεδρία. Ήταν θαυμάσια αυτή η συνεργασία που επέτρεψε τα αποτελέσματα αυτά, τα οποία ήταν απαραίτητα, αλλά και κατεπηγόντως απαραίτητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κρίσει τροφοδοσία είναι, είναι πολύ συχνέ δυστυχώ και αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο για πολλέ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στην οικονομία και την ανταγωνιστικότητα των χωρών αυτών. Αυτή η έκθεση λοιπόν είναι ένα σημαντικό βήμα στο να μπορέσει να επιτευχθεί μια σειρά στόχων που έχουμε θέσει ως Ευρωπαίοι για την ασφάλεια εφοδιασμού σε λογικές τιμές και με έναν τρόπο που σέβεται το περιβάλλον. Τα συμπεφωνημένα μέτρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικά και έχουν επιτευχθεί συμφωνίες ουσιαστικές οι οποίες δείχνουν και το μεγάλο ταλέντο διαπραγματευτικό του κ. Βιδάλ Κουάντας. Θέλω να τον ευχαριστήσω και πάλι λοιπόν κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ λέει και ο Πρόεδρος. Ερχόμαστε είμαστε στο τέλος του σημείου αυτού της ημέρησης διάταξης και ελπίζουμε ότι θα έχουμε και την ευκαιρία να το αποφασίσει πλήρως το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα τώρα να, να χαιρετήσω τον κύριο Φελίπε Πέδρες Γάλμπο, ο οποίος είναι ο υφυπουργό για τα θέματα βιομηχανίας έρευνας και ενέργειας, εκπροσωπεί την ε, Υπουργό κυρία Κάρμεν Γκάρμεντία η οποία δεν μπόρεσε να είναι παρούσα σήμερα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας. Έχετε το λόγο. Και έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Ήτρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα καταρχήν να σας ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση στην έλευσή μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή σας, διότι μια απεργία των ελαγκτών ενέργειας κυκλοφορίας με καθυστέρησε περίπου δύο ώρες και φυσικά θέλω να ζητήσω και συγγνώμη εξ ονόματος της κυρίας Γκαρμεντία, η οποία δεν μπόρεσε να είναι παρούσα σήμερα, όπως θα είχε σίγουρα θελήσει, διότι έχει προσκληθεί σε μια, έχει προσκληθεί σε μια πάρα πολύ σημαντική συνεδρίαση στην Ισπανία όπου πρέπει να είναι παρούσα. Είναι λοιπόν μια μεγάλη χαρά για μένα που μπορώ να ευχαριστώ ενώπιόν σα για να σα παρουσιάσω τα αποτελέσματα και τον απολογισμό τη Ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου στα θέματα έρευνας. Στις 28 Ιανουαρίου η κυρία Καρμεντία ήταν ενώπιόν σα και τότε είχε μόλις αναλάβει η Ισπανία την Προεδρία του Συμβουλίου έρευνα σε μια στιγμή η οποία ήταν κομβική για το θεσμικό και πολιτικό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια νέα συνθήκη, με μια νέα κομισιόν που δεν είχε ακόμα εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη στρατηγική 2020 η οποία ακόμα δεν είχε καθοριστεί πλήρως και με μια πλήρη ημερήσια διάταξη για θέματα που αφορούσαν το Συμβούλιο ε, Ανταγωνιστικότητας μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται και η έρευνα. Πέραν του θεσμικού πλαισίου το οικονομικό και χρηματοοικονομικό στερέωμα ήταν και εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολύπλοκο. Παρά τις δυσκολίες αυτές, εμείς στοχεύσαμε να έχουμε μια δυναμική και φιλόδοξη Προεδρία που δεν ήθελε να αποχωριστεί κανένα από τους αρχικούς της στόχους. Για την επίτευξη αυτών των στόχων προχωρήσαμε σε ένα δυναμικό και έντονο πρόγραμμα με προτεραιότητες οι οποίες καθορίζονται από τους τρεις βασικούς άξονές μας, η ενσωμάτωση, η συμμετοχή και η περιεκτικότητα. Για μας η ενσωμάτωση και η ολοκλήρωση σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε σημασία στις πολιτικές έρευνας και ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, ώστε ο Ευρωπαϊκός χώρος ε, έρευνας, ΕΡΑ, να συμμετέχει πλήρως και να ενσωματώνεται σε όλες τις πολιτικές καινοτομίες, ιδίως στην πολιτική της ε, επίτευξης των στόχων του 2020 και των στόχων των κρατών μελών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τη ενσωμάτωση έχουμε προχωρήσει σε σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με τη διακυβέρνηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνα, με την τροποποίηση των δομών και μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνα, του ERC, και με την τύποση αυτών των στόχων για, για να έχει και η Τεχνική και, και Επιστημονική Επιτροπή μεγαλύτερο πολιτικό βάρος αυτή η επιτροπή, η οποία έχει τώρα τον τίτλο Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνα, θα συμμετέχει ακόμα περισσότερο σε ό,τι αφορά τη χάραξη κοινών στόχων για την ευρωπαϊκή έρευνα. Συγχρόνω, κάναμε ένα σημαντικό βήμα για μια Ευρώπη ολοκληρωμένη γνώση, για να αντιμετωπίζοντα την κινητικότητα και την επαγγελματική καριέρα των Ευρωπαίων ε, ερευνητών στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα του Μαρτίου. Παρουσιάσαμε συνέχεια τα συμπεράσματά μα για πρώτη φορά στο Συμβουλίο Κοινωνικών Θεμάτων Υγείας και Καταναλωτών. Θεωρούμε ότι αυτό ήταν πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να θεσπίσουμε μια πέμπτη ελευθερία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ελευθερία κυκλοφορίας των γνώσεων και της πληροφορίας. Τονίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία έτυχε πολύ θετική αποδοχή και από το Συμβούλιο των Υπουργών και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό της στρατηγικής της Ευρώπης 2020, Θέλω να τονίσω ότι και τα, τα δύο συμβούλια ανταγωνιστικότητας που έχουν λάβει χώρα, όπως και στην άτυπη σύνοδα του Φεβρουαρίου, αντιμετωπιστήκαν ορισμένα από τα θέματα της στρατηγικής αυτής και φυσικά αυτή η στρατηγική περιλαμβάνει στόχους και ενδείκτες που έχουν οικοδομηθεί επί τη βάση του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας. Έγινε σαφής επίσης η ανάγκη να περιλάβουμε δείκτες οι οποίοι αντανακλούν τις εκτιμήσεις σε σχέση με τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της έρευνας και ανάπτυξης. Θεωρούμε ότι ο νέος αυτός στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να υπάρξει μεγαλύτερη <clears throat> επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη και που θα εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο, αντανακλά αυτή την αντιμετώπιση. Για να υπάρξει ένα πιο ολοκληρωμένο χώρο έρευνα επίση, έχουμε αντιμετωπίσει σημαντικά θέματα όπω η επιστημονικές υποδομές που περιλαμβάνονται στον ε, οδικό χάρτη των μεγάλων υποδομών για την σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, για την υποστήριξη των γυναικών στην ε, επιστήμη και, της ευρωπαϊκή, και τεχνολογία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα θέματα αυτά περιλαμβάνονται σε συμπεράσματα που ενεκρίθησαν το Συμβούλιο για διάφορες πτυχές του ευρωπαϊκού ερευνητικού χώρου. Επίσης, σε ό,τι αφορά τον άξονα αυτό της ολοκλήρωσης, η Ισπανική Προεδρία ε, προέτεινε κατευθύνσει στο Συμβούλιο που έγιναν δεκτές σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο θα διατυπωθεί το επόμενο ε, Ευρωπαϊκό Σχέδιο καινοτομία και έρευνα που ελπίζω θα παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο. Θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο να συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε για το πώ θα δημιουργήσουμε μια καινοτόμα Ευρώπη, Ευρώπη για να προχωρήσουμε σε ορισμένα σημεία τα οποία από την ειδική μας οπτική γωνία είναι πάρα πολύ σημαντικά να τα εξετάσει και η Κομισιόν. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου αρθρώνονται σε πέντε κύριους άξονες, χρηματοδότηση, αγορές, διακυβέρνηση, περιφέρειες και άτομα. Σε σχέση με το δεύτερο άξονα της Ισπανικής Προεδρίας, της ε, συμμετοχής, θεωρούμε ότι τα προγράμματα αυτά έρευνας και κοινοτομίας, είτε είναι κοινοτικού χαρακτήρα εθνικά ή διακυβερνητικά, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και τις μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Νέες πηγές ενέργειας και κλιματική αλλαγή, γύρανση του πληθυσμού και ασθένειες, οικονομική κρίση. Θεωρούμε επίση ότι αυτή η απάντηση που θα δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι αποτελεσματική να οδηγήσει σε απλοποίηση του έργου των ερευνητών και ακολουθώντα αυτή την οδηγό γραμμή. Θέλω να τονίσω ότι το κύριο θέμα το οποίο έθιξε η Προεδρία μα κατά τη διάρκεια τη άτυπη Συνοδού των Υπουργών ε, έρευνας που έγινε στο Σαν Σεμπάστιαν στις 8 Φεβρουαρίου ήταν η λεγόμενη δήλωση του Σαν Σεμπάστιαν τον Όστια με τίτλο «Η επιστήμη για την ανάκτηση της οικονομικής ανάκαμψης εδώ και τώρα». Αυτό το έγγραφο που υποστηρίχθηκε ομόφωνα από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τονίζει το ρόλο που μπορεί να έχει η επιστήμη για να δώσει απαντήσεις και λύσεις που θα οδηγήσουν στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Για να μπορέσει λοιπόν <clears throat> να υπάρξει πλήρης παρουσία και συμμετοχή της έρευνας και της καινοτομία στις πολιτικές μας, πρέπει να υπάρχει και καλύτερη πρόσβαση στα ευρωπαϊκά προγράμματα, που θα πρέπει να είναι πιο απλά και πιο αποτελεσματικά. Όπως γνωρίζετε, η απλοποίηση είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει τύχει μεγάλη προτεραιότητα για την Ισπανική Προεδρία και είναι κάτι το οποίο πάντα επανέρχεται για το Συμβούλιο όταν συζητούμε για θέματα έρευνας. Είναι απαραίτητο και για την ε, ε, για όλους τους κοινωτικούς θεσμούς και για όλους τους φορείς που συμμετέχουν στα προγράμματα πλαίσιο και ιδίω αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την αντιμετώπιση τους. Θεωρεί ο Προεδρία ότι είναι μια απαράγραπτη προϋπόθεση η απλοποίηση για την οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνα και για τη στρατηγική του 2020 ευρεία τη έννοια. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια απλοποίηση των διαδικασιών και των προτύπων και να υπάρξει μια μετατόπιση παραδείγματος η οποία θα επιτρέψει να περάσουμε σε ένα σύστημα που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και όπου το σημαντικό είναι να δοθεί προτεραιότητα σε μια έρευνα ποιότητα και τη οποία η χρηματοδότηση να βασίζεται στα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Ιδίω για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει θεωρούμε ότι αυτέ οι αλλαγέ θα είναι θετικέ και θα του επιτρέψουμε να βελτιστοποιήσουν τι προσπάθειέ του και να συγκεντρώσουν καλύτερα του πόρου του στην έρευνα και να μειώσουν επομένω και το διοικητικό άκθο που επομίζονται. Αυτή ήταν λοιπόν η άποψη της, Ισπανική της Ισπανικής Προεδρίας και για μας ήταν μεγάλη χαρά το, ότι μπορέσαμε να προωθήσουμε την έγκριση σημαντικών ε, συμπερασμάτων στο Συμβούλιο του Μαΐου για τα θέματα αυτά. Συγχρόνως, αυτό είναι αλληλένδετο με την κοινωνική διάσταση του ευρωπαϊκού ε, ερευνητικού χώρου. Και έρχομαι τώρα στον τρίτο άξονα της δράσης μας, που είναι η συμπερίληψη. Θεωρούμε λοιπόν ότι η έρευνα και η καινοτομία θα πρέπει να έχουν ένα μεγαλύτερο ρόλο στον αγώνα κατά της ένδυας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η Ισπανική Προεδρία θεωρεί ότι η γνώση, η Ευρώπη της γνώσης θα πρέπει να οδηγεί προς μια στρατευμένη επιστήμη και με μεγαλύτερη ευαισθησία για αυτά τα κοινωνικά θέματα. Θεωρήσαμε ότι πρέπει να συμπληρωθούν τα οράματά μας σε σχέση με, τους, με τις μεγάλες προκλήσεις που έθεσε η Σουηδική Προεδρία και να συνεχίσουμε τις δράσεις μας κατά της ένδυας και της ανισότητος γιατί είναι και ένας από, τους, από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την επιστήμη μας. Η Προεδρία θέλει να προωθήσει λοιπόν αυτή τη δήλωση αυτή την πρωτοβουλία, δέκα χρόνια μετά τη δήλωση των στόχων της χιλιετίας, μετά από τη στρατηγική Λισαβόνας και μέσα στο ευρωπαϊκό έτος κατά της ένδυας και του κοινωνικού αποκλεισμού για να χρησιμοποιήσει το τεράστιο δυναμικό της έρευνας και της τεχνολογίας για να έχουμε και την ανθρώπινη ανάπτυξη και όχι μόνο η οικονομική ανάπτυξη. Με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαΐου έχει δοθεί έμφαση για πρώτη φορά στη σημασία της ανάπτυξης της κοινωνικής διάστασης του ευρωπαϊκού ερευνητικού χώρου ως εγκάσιας μεθόδου προώθησης της αριστείας σε τεχνολογικό και επιστημονικό χώρο και διερεύνησης κοινού χώρου μεταξύ της ε, ανάπτυξης, της συνεργασίας για την ανάπτυξη και της έρευνας και ανάπτυξης και συγχρόνως μειώνοντας την ένδια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Και αυτό συνάπτεται άμεσα με τη στρατηγική της Ευρώπης του 2020 και επίσης με το στόχο κατά προτεραιότητα της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Από νομοθετική έποψη η Ισπανική Προεδρία είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη γιατί κατάφερε να διεκπαιρεώσει πλήρω δύο πρωτοβουλίε στο πλαίσιο τη Νέα συνθήκη τη Λισαβόνα και σε πλαίσιο συναπόφαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για την απόφαση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου σε σχέση με τη συμμετοχή τη της Ευρωπαϊκής στο κοινό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης για τη Βαλτική θάλασσα, τον Πόνου 169, με παρουσία πολλών κρατών μελών και επίσης η έγκριση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε σχέση με το πρόγραμμα ε, παρακολούθησης της γης και τις αρχικές δράσεις στον τομέα αυτό 2011-2013. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την καρποφόρα συνεργασία μεταξύ των θεσμικών αυτών οργάνων καθ' όλη τη διάρκεια έγκριση αυτών των, των ε, προτάσεων και για το θαυμάσιο έργο των δύο εισηγητών της Λένα Εκ και του Νόρμπερ Γκλάντερ που έχουν συμβάλει με ουσιαστικό τρόπο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος εξαμήνου, το Υπουργείο Έρευνας <clears throat> και Επιστήμης, όπως σας είπα, συγκάλεσε μια άτυπη συνεδρίαση υπουργών στο Σαν Σεμπαστιάν Ντονοστία και δύο συμβούλια ανταγωνιστικότητας, τα οποία μπορέσαμε να καταλήξουμε σε ευρωπαϊκή συνένεση για πάνω από 30 ζητήματα στην πολιτική ε, ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης και 40 εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Προεδρία και τα Υπουργεία της. Θεωρούμε ότι η Ευρώπη της Συνθήκης Λισαβόνας θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη φωνή στους πολίτες και εμείς ως Προεδρία προσπαθήσαμε να προωθήσουμε κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να τονίσω ότι χάρη στη σημαντική συμμετοχή και το ενδιαφέρον και το υψηλό περιεχόμενο των εκδηλώσεων που οργάνωσε η Ισπανική Προεδρία κατέστη να τον επιτρέψουμε στους κυρίους εμπλεκομένους <clears throat> στους τομείς της έρευνας και της καινοτομία να συμβάλλουν μέσα και από τα, από τα συμπεράσματα των εκδηλώσεων αυτών σε μια σημαντική προώθηση στα ζητήματα αυτά που αντιμετωπίσαν τα Συμβούλια ανταγωνιστικότητα κατά διάρκεια του εξαμήνου τη Προεδρία μα. Θέλω επίση να αναφέρω <clears throat> ότι η Ισπανική Προεδρία κατέβαλε μια ιδιαίτερη προσπάθεια και πιστεύουμε ότι συνέβαλε σημαντικά για να μπορέσει να επιτευχθεί μια ευρωπαϊκού χαρακτήρα συνένεση σε σχέση με την χρηματοοικονομική βιωσιμότητα του ε, μεγάλου διεθνούς προγράμματος ΙΤΕΡ για τη θερμοπυρηνική σύνδεξη. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας την παρέμβασή μου, <clears throat> όπως σας έλεγα στην αρχή, γνωρίζαμε ήδη εν τη ενάρξη της Προεδρίας μας ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε σημαντικές προκλήσεις, αλλά όχι προκλήσεις που θα ήταν αδύνατο να αντιμετωπίσουμε. Διότι ήταν και η στιγμή της ε, κύρωσης της συνθήκης Λισαβόνας και της ανάληψης εξουσίας της νέας Κομισιόν. Συνεχίζουμε να είμαστε δυναμικοί και φιλόδοξοι για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε προόδους στην Ευρώπη της ε, πληροφορίας και της γνώσης. Χωρίς να ξεχνούμε το σήμερα και χωρίς να ξεχνούμε τις ανάγκες της Ευρώπης υπέρ των πολιτών μιας Ευρώπης η οποία διέρχεται δύσκολες οικονομικές ατραπούς. Και εν συμπεράσματι και επί τη βάση της δικής μας Κατεύθυνση προς την ενσωμάτωση, τη συμμετοχή και τη συμπερίληψη, είμαστε πεπισμένοι ότι συμβάλλουμε σημαντικά για την περαιτέρω ανάπτυξη του χώρου έρευνας της Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη βελτίωση συγκεκριμένων στοιχείων της Ευρωπαϊκής Έρευνας που σε ορισμένε περιπτώσεις για πρώτη φορά έχουν τεθεί στην ημερησία διάταξη της Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι για μένα λοιπόν μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση το γεγονός ότι μπορώ να τονίσω ενώπιόν σας ότι η Ισπανική Προεδρία έχει αναπτύξει πλήρως και έχει επιτύχει όλους τους στόχους και την πολιτική ατζέντα που έθεσε στην αρχή του εξαμήνου αυτού συγχρόνως και έχει διοργανώσει μια μεγάλη σειρά από διασκέψεις και εκδηλώσεις. Θέλω παρόλα αυτά να τονίσω ότι η έρευνα και η επιστήμη καθώς και η καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν να αντιμετωπίσουν ακόμα σημαντικές προκλήσεις, πολλές από τις οποίες είναι απόρριε τη δύσκολη οικονομική και χρηματοοικονομική κατάσταση σε διεθνέ επίπεδο και επίση από την ανάγκη των κρατών μελών να αποφασίσουν πώ θα χρησιμοποιήσουν του ισχνού δημόσιου πόρου του που βρίσκονται κάτω από μεγάλη πίεση για τι περισσότερε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό οι χώρε μα να συνεχίσουν ακόμα και στο μέλλον να επενδύουν σημαντικά ποσά στην καινοτομία και στην έρευνα και ανάπτυξη. Γι' αυτό θέλω να τονίσω τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζετε όλοι σας <clears throat> ως μέλη ενός θεσμού όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που παίζει σήμερα ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στις πολλές αποφάσεις οι οποίες αφορούν τον κοινοτικό προϋπολογισμό για τα επόμενα χρόνια. Είναι απαραίτητο το όραμα αυτό της Ευρώπης του σήμερα και του αύριο που ελπίζω ότι είναι ένα κοινό όραμα να μπορέσει να γίνει κατανοητό και να υποστηθεί και από τους Ευρωπαίους πολίτες που είναι τελικά ο απότερος αποδέκτης και ο λόγος ύπαρξης όλων των πολιτικών μας και είναι ο, οι πολίτες αυτοί στους οποίους εμείς είμαστε υπόλογοι. Γι' αυτό είναι σημαντικό και εσείς από τη δική σας θέση να υποστηρίξετε στεναρά την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της να μην ξεχάσουν το σημαντικό αυτό στίχημα της, έρευνα, της έρευνας ανάπτυξης και καινοτομίας. Επειδή αυτή είναι μια από τις τελευταίες παρουσίες μου Εκ ονόματος τη Ισπανικής Προεδρίας θέλω να, να τονίσω την σημασία της συνεργασίας σας και να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη συνεργασία σας και θέλω να διαβιβάσω στο Βέλιο και την Ουγγαρία της επερχόμενης προεδρίας όλη την υποστήριξή μας για το δύσκολο αυτό έργο που έχουν να αντιμετωπίσουν. Πιστεύω επίση ότι είναι απαραίτητο να ευχαριστήσω δημόσια όλη την ε, ομάδα της Ισπανικής Προεδρίας που χάρη στην παρουσία της και τις προσπάθειές της ε, μας έδωσε τη δυνατότητα να επιτύχουμε όλους αυτούς τους στόχους της Ισπανικής Προεδρίας και θέλω και πάλι εκ βάθους καρδίας να τους ευχαριστήσω για την επιτεύξη αυτών των στόχων που διατυπώσαμε στην αρχή του έτους. Προφανώς παραμένω στη διάθεσή σας για τα ερωτήματα τα οποία θέλετε θέση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και την παρουσία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, τη σύνοψη και για τη συνεργασία. Κάποιοι συνάδελφοι ζήτησαν ήδη το λόγο. Πρώτα απ' όλα η κυρία Ρέιρα Μαδουρέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα κύριε Υφυπουργέ να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας ενώπιον της Επιτροπής μας και να σας συγχαρώ εξ ονόματος της ομάδας μου για το έργο το οποίο έκανε και το Υπουργείο Έρευνας Επιστήμης μάλλον και καινοτομία σε αυτό το εξάμεινο. Νομίζω το έχετε εξηγήσει πολύ καλά ότι υπήρξε αυτή η εργόδης και έντονη προσπάθεια να ευοδοθεί το πρόγραμμα εργασίας το οποίο ήταν πλήρες και φιλόδοξο όπως μας το παρουσίασε η κυρία Γκαρμενδία στην αρχή της του εξαμήνου της Ισπανικής Προεδρίας, ένα πρόγραμμα το οποίο συνάδει με τις ανησυχίες και τους στόχους της δικής μας Επιτροπής και χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι στο μεγαλύτερο μέρος του αυτό το πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ιδιαίτερα τις πρόοδους οι οποίες επετέφθησαν σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου έρευνα. Στους τρεις άξονες που αναφέρατε, κινητικότητα, δείκτες, υποδομή και όλα αυτά. Υπήρξαν σημαντικές πρόοδοι. Θέλω όμως να υπογραμμίσω ιδιαίτερα το γεγονός ότι για πρώτη φορά στα, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου έχει δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και να σας συγχαρούμε ιδιαίτερα για αυτό. Βέβαια, το δύσκολο να περάσει κανείς από τη θεωρία στην πράξη. Και σε αυτό το σημείο στρέφεται και το ερώτημά μου. Στην πράξη, πώς προσδοκείτε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σε σχέση με την κοινωνική διάσταση του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Χώρου να αντανακλώνται στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και ένα δεύτερο θέμα το οποίο πηγαίνει προς την ίδια κατεύθυνση, οι πολιτικές κατευθύνσεις της Ισπανικής Προεδρίας σε σχέση με την καινοτομία, πώς θα υλοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο είτε, είτε κοινοτικό είτε διακυβερνητικό και τέλος θέλω να σας συγχαρώ για όλα αυτά τα μέτρα τα οποία προωθήσατε για να υπάρχει μια πιο ισορροπημένη παρουσία μεταξύ ανδρών και γυναικών στον επιστημονικό και τεχνολογικό χώρο, ώστε να χρησιμοποιήσουμε όλο το δυναμικό μας ως Ευρώπη και όχι μοναχά το μισό. Αυτό είναι κάτι το κεφαλαιόδες για να μπορέσουμε <clears throat> όχι μόνο να είμαστε συνεκτικοί με τις ευρωπαϊκές μας αξίες, αλλά και για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους ανταγωνιστικότητάς μας. Αυτά και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Χέρτσογκ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Υφυπουργέ, λίγα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στην Ισπανική Προεδρία όταν ξεκίνησε η κρίση νόμιζα πως θα έρχεται όλο το βάρος στις χρηματαγορές. Έγινε μια ιδιαίτερη προσπάθεια να παραμείνει η έρευνα καινοτομία στην κορυφή όταν όλοι μιλούσαν για τα λεφτά. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για αυτά τα οποία επιτύχατε και για τη στρατηγική 2020 και για το GMS και, την... και τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Θα ήθελα επίσης να σας συγχαρώ για την ομάδα που έχετε εδώ πέρα στις Βρυξέλλες γιατί συνεργαστήκαν πάρα πολύ σε αυτές τις πολιτικές. Θα ήθελα να κάνω και μια ερώτηση για τα δημοσιονομικά μέσα για το πώς θα επιτύχουμε τα, της πολιτικής Λισαβόνας όπως πολιτική του διαστήματος, η ΤΕΡ κτλ. Η Επιτροπή μας, ξέρετε, είναι βιομηχανίας και έρευνας και δεν θα θέλαμε να κοπούν έργα του πρόγραμματος πλαισίου 7 επειδή δεν έχουμε προϋπολογισμό. Πρέπει να σώσουμε το πρόγραμμα πλαισίου 7. Θα ήθελα να καταλάβει το Συμβούλιο πως αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε δεν είναι πρόκληση προϋπολογισμού, είναι πρόκληση δημοκρατική. Υπονομεύουμε τις νέες ικανότητες Λισαβόνας να τα κάνουμε αυτά. Θα έχετε λοιπόν το κουράγιο να σπάσετε την ηγεμονία του ΕΚΟΦΗΝ και να μην τους επιτρέπετε να κόψουν ε, τους δημοκρατικούς στόχους ε, που έχουμε θέσει λόγω έλλειψης ε, χρημάτων. Ευχαριστώ και εμείς θα σας βοηθήσουμε οπωσδήποτε αν κάνετε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Λάγιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Φιβουργέ. στις 3 Μαρτίου στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας ε, το Συμβούλιο μετά από δική σας ε, πρωτοβουλία ξεκαθάρισε πως θα πρέπει να υπάρξει μια βιομηχανική πολιτική και ζήτησε από την Κομισιόν να προετοιμάσει μια ανακοίνωση την οποία προετοιμάζει η Κομισιόν. Ίσως θα μπορούσατε λοιπόν να μας πείτε από τη δική σας σκοπιά ποια στοιχεία βλέπετε όσον αφορά την καινοτομία να περιέχονται σε μια τέτοια ανακοίνωση για τη βιομηχανική πολιτική του μέλλοντος. Ποια συνεισφορά βλέπετε από την σκοπιά της έρευνας και της καινοτομίας για μια τέτοια βιομηχανική πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νίστελ Ρόι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εμείς στο ΕΛΚ έχουμε θετική εντύπωση από αυτά τα οποία έχετε κάνει. Επικεντρωθήκατε στο κομμάτι της ανταγωνιστικότητας και στο ρόλο που παίζει η έρευνα. Ενδιαφέρον είναι που είπατε πως ε, θα δείτε τώρα θα γίνει με τη Βελγική Προεδρία Ποια είναι τα πιο κρίσιμα ζητήματα για σας όσον αφορά τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνα στη διακυβέρνησή του και τι πρέπει να γίνει να ολοκληρωθεί τους ερχόμενους μήνες. Δεύτερον, είχε πάρα πολλές ε, ε, δραστηριότητες στο Συμβούλιο, Συμβούλια επίσημα και άτυπα. Υπήρχε αυτή η εβδομάδα για τις καινοτόμες ε, περιφέρειες ε, στη Σαραγώσα με 500 συμμετέχοντες από περιφέρειες, πανεπιστήμια, πόλεις κτλ. Το ερώτημά μου είναι, αναφέρατε την κοινωνική διάσταση, Αλλά εδώ στο Κοινοβούλιο ε, είδαμε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε και συνέργεια στα ταμεία και με την κοινωνική διάσταση. Αλλά υπάρχει περιφερειακή διάσταση. Κάτι το οποίο είναι καινούριο στη συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Οπότε δεν θα πρέπει μόνο να έχουμε έξυπνους ερευνητές που θα ταξιδεύουν ελεύθερα, αλλά να υπάρχει και κάπου ένας χώρος που θα γίνεται αυτή η έρευνα, κάποιοι πόλη εξειδίκευσης. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω τι πρόοδο βλέπετε σε αυτό, δηλαδή η συνέργεια μεταξύ των διαφόρων ταμείων και ποια θα μπορέσει να είναι η εξειδίκευση η τοπική στις διάφορες περιφέρειες. Σας ευχαριστώ, Μπέιβερ. Υπουργέ, η Ισπανική Προεδρία υπογράμμισε και όλοι χαίρονται γι' αυτό την ανάπτυξη της έρευνας, την ανάπτυξη, την καινοτονία στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ ο ίδιος είμαι αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας ε, μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και βλέπω πόσο γρήγορα οι αναδυόμενες χώρες προσπαθούν να αναρριχηθούν και αυτές, να δια να κάνουν πρόοδο στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Βλέπω στην Ινδία και σε άλλες χώρες ε, τι γίνεται και νομίζω ότι στριμωχνόμαστε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών που εξακολουθούν την μεγάλη τους κούρσα προς τα μπροστά, τον αγώνα δρόμου τους και μεταξύ των άλλων αναδυόμενων δυνάμεων που αναπτύσσονται ταχύτατα. Όπως ξέρετε, στην Ινδία παράγονται 300.000 ε, ειδικοί πληροφοριών και μηχανικοί ε, και ειδικοί όχι μόνο στην ε, έρευνα αλλά και υπάρχει και μετατόπιση των τμήματων έρευνας και τεχνολογίας των επιχειρήσεων προς αυτές τις χώρες. Χαίρομαι πολύ που αντιμετωπίζετε με προσοχή αυτό το φάκελο και ελπίζω ότι και οι διάδοχοί σας θα διπλασιάσουν ακόμα περισσότερο τις προσπάθειές τους πρέπει να προσθέσω μια ερώτηση στις ερωτήσεις των συναδέλφων. Τι έχουμε κάνει, τι πρόοδος έχει σημειωθεί, τι μπορούμε να ελπίζουμε στον τομέα των Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, που είναι μία από τις ασχήλιες πτέρνες ε, της ε, δραστηριότητάς μας στον τομέα αυτό. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ, Υπουργέ. Ε, οι συνάδελφοι ανέφεραν πολλά πράγματα. Τις τελευταίες 6 με 8 μήνες, μια χώρα που έχει αντιμετωπίσει τόσο σοβαρή κρίση και κατάφερε να φέρει σε πέρα στην Ευρωπαϊκή Προεδρία ε, πραγματικά εκτιμούμε τις ικανότητες και τις προσπάθειές σας. Ε, προσπαθήσατε να έχετε πάντοτε στο προσκήνιο την ευρωπαϊκή ιδέα ε, και με επιτυχία κρατήσατε τα ενία της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Συγχαρητήρια για τις προσπάθειές σας. Έχω δύο ερωτήσεις που συνδέονται μεταξύ έρευνας και επιστήμης. Ξέρω ότι επειδή είστε ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες σε τεχνολογίες όπως η συγκεντρωμένη ηλιακή, συγκέντρωση ηλικής δύναμης, η αιωλική ενέργεια και άλλες, πραγματικά προσπαθήσατε να σημειώσετε πρόοδο στο κρίσιμο ζήτημα που είναι η χρηματοδότηση όλων αυτών των πραγμάτων. Ξέρουμε ότι είναι ένα δύσκολο θέμα. Κανείς δεν έχει μια εύκολη απάντηση. Ύστερα από, αυτές τις έξι, από αυτούς τους έξι μήνες, ίσως θα μπορούσατε να μας δώσετε δύο-τρεις ιδέες ε, για το πώς μπορούμε να συνεχίσουμε ε, εν ώψη και των δημοσιονομικών προοκτικών, με τα εισοδήματα που θα έχουμε από το διοξίδιο του άνθρακα και από τον εκπληστηριασμό των σχετικών δικαιωμάτων. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε με αυτά. Επίσης, ε, νομίζω ότι κληρονομήσατε πολύ δύσκολα θέματα. Το θέμα της χρηματοδότησης ε, του πυρηνικού αντιδραστήρα. Το λεγόμενο ITER. Έχετε κάποιες ιδέες ε, Πού θα βρούμε αυτά το 1,5 ή 1,4 εκατομμύρια ευρώ που θα χρειαστούμε μέχρι το 2012 και 2013. Βασικά άκουσα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο ενός δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ξέρω με επαφές που έχω με την γερμανική κυβέρνηση ότι η Γερμανία δεν θα το δεχτεί αυτό, δεν θα δεχτεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ένα δάνειο από το οποίο δεν θα αναμένει κάποια ιδιαίτερη απόδοση. Επίσης, άλλο άλλη μια επιλογή είναι περισσότεροι πόροι από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Έχετε συγκεκριμένες ιδέες. Η κυρία Χέρτσοκ ήδη το ανέφερε. 1,4 δισεκατομμύρια πρέπει να προέλθουν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό μέχρι το 2012-2013. Πώς θα το κάνουμε όμως αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω, είσαστε υπέρ και του προγράμματος Γαλιλαίος ε, από ό,τι κατάλαβα, ήδη κάνατε μια, δώσατε μια πολύ εύγλωτη ομιλία για την ε, σημασία της ευρωπαϊκής έρευνας. Από πού θα προέλθουν όλα αυτά τα χρήματα. Από ποιες περικοπές, ε, από ποια κατανομή του κοινοτικού προϋπολογισμού θα προέλθει αυτό το 1,4 εκατομμύριο ευρώ, γιατί αυτό χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ κύριε Υπουργέ θα ήθελα <clears throat> να, να σας πω ότι έχετε καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ως Ισπανική Προεδρία. Ο απολογισμός σας είναι ιδιαίτερα θετικός. Ήταν ένα από τα πιο καρποφόρα προγράμματα εργασίας εξάμενης προεδρίας και θέλω να σας θέσω ένα πάρα πολύ σύντομο ερώτημα το οποίο είχα ήδη απευθύνει ε, και στο παρελθόν στα πλαίσια των εργασιών της Επιτροπής μας με τις στρατηγικέ καινοτομίε. είναι το ερώτημα και έρευνας που έχετε αναπτύξει <clears throat> σε σχέση με την μελλοντική τώρα χρηματοδότηση αυτών των ενεργειών θα ήταν χρήσιμο να προβλέψουμε να έχουμε λοιπόν μια συνεργασία και σε επίπεδο κρατών μελών για καλύτερη συμμετοχή στην ε, χρηματοδότηση αυτών των ενεργειών ώστε να υπάρχει μια προσαρμογή στις ανάγκες αυτών των κρατών. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Υπήρξε ένα, μια πλειάς ερωτήσεων που σας έχει απευθυνθεί, κύριε Υφυπουργέ, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να δώσετε απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Ε, lugar... Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι έλαβαν το λόγο. Να σε ευχαριστήσω για αυτό που είπατε και για το πώς το είπατε. Για μας ήταν μια μεγάλη ικανοποίηση να μπορέσουμε να ηγηθούμε, να κρατήσουμε το πιδάλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την έρευνα και την ανάπτυξη αλλά και την καινοτομία. Επομένως, καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω. Κάποιοι από τους ομιλητές έθεσαν ζητήματα τα οποία λίγο πολύ επικαλύπτονται. Ε, θέλω να απαντήσω με κάποιες πρώτες σκέψεις ακολουθώντας τη σειρά των ερωτημάτων που τέθηκαν. Βέβαια, αν χρειάζεται άλλες πληροφορίες, είμαι πάντα στη διάθεσή σας, όπως και οι υπηρεσίες μου. <clears throat> Ξεκινώ λοιπόν στην κυρία Ρίαρα Μαδουέλ, η οποία αναφέρθηκε όλος ιδιαίτερος στις πρόοδους οι οποίες έχουν επιτευχθεί για τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνα και συγκεκριμένα για δύο σημεία. Καταρχήν το θέμα της κοινωνικής ε, διάστασης του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας, το οποίο αναφέρθηκα και εγώ ίδιος. Εδώ υπάρχει και το ίδιο το πάθος για την έρευνα, όταν η έρευνα έχει κοινωνικά αποτελέσματα, κοινωνικό αντίκτυπο. Πρέπει να διέπεται η έρευνα από την αρχή της κοινωνικής ευθύνης για να μπορούμε να είμαστε επιτυχείς σε ό,τι αφορά την διάσταση αυτή θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε και οι πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα τις προσπάθειές μας και αυτό θα ενισχύσει το σύνολο σύστημα. Μπορούμε λοιπόν σίγουρα να συμφωνήσουμε για τις αρχές. Έχει φτάσει τώρα η στιγμή, και το έμαθα από την κυρία Καρμενδία, πρέπει να περάσουμε τώρα από τα λόγια στην πράξη και να καλύψουμε τα θέματα κοινωνικής δέσμευσης και στράτευσης που είναι πολύ πιο εύκολο εδώ να υπάρχει συμφωνία στα λόγια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όμως να υλοποιήσουμε τις απαραίτητες πολιτικές και αυτό φαίνεται στα εμπόδια που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. <clears throat> Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τις αρχές αυτές και στην υλοποίηση των των πολιτικών μας. Αλλά νομίζω ότι με τις ε, συστάσεις, τις προτάσεις που μας έγιναν, έχουμε καταλήξει σε μια σειρά συμφωνίων για να υποστηρίξουμε ιδιαίτερα περιπτώσεις που θίγεται η έρευνα από την οικονομική κρίση. Εμείς θα πρέπει καταρχήν να προωθήσουμε τη μεγαλύτερη προσβασιμότητα των πολιτών στην ε, επιστημονική και τεχνολογική δραστηριότητα. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ για το γεγονός ότι συμμετέσχουν χίλιοι περίπου πολίτες σε μια εκδήλωση η οποία οδήγησε στην ε, προτάσεις επιλογής ε, σχεδίων και προγραμμάτων για την έρευνα. είναι μια ένδειξη του τι θέλουν οι πολίτες. Θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία να μπορούμε να ακούσουμε τις απόψεις τους και να ξέρουμε ότι αυτές είναι οι προτάσεις τους και πρέπει να ληφθούν υπόψη και αυτό σημαίνει βέβαια και μια μεγαλύτερη συμμετοχή σε θέματα όπως είναι η υδροδότηση, η υγεία, η παιδεία κτλ. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη γιατί είναι ιδιαίτερα προσφυλή στους πολίτες. Δεύτερο ερώτημα. Προσπαθώ να είμαι σύντομος βέβαια, δεν ξέρω αν μακρύγορο ιδιαίτερα. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η πρόθεση των πολιτικών καινοτομία. Το σχέδιο αυτό έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομία, το οποίο νομίζω ότι την χάνει απόλυτη σύμνοια όλων. Έχει εργαστεί προς την κατεύθυνση αυτή η Ισπανική Προεδρία επί τη βάση των πέντε αυτών αξώνων που σας ανέφερα προηγουμένως. Το ερώτημα είναι πώς θα υλοποιηθούν αυτά στα κράτη-μέλη. Και εδώ θα πρέπει εγώ να αναφερθώ στην περίπτωση της Ισπανίας που ξέρω καλύτερα. Παράλληλα με τις πολιτικές προώθησης της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας μάλλον, προχωρήσαμε και στην στρατηγική καινοτομία μέσα στο έδαφος της Ισπανίας. Ένα σύνολο λοιπόν <clears throat> δραστηριοτήτων για το 2010 και προβλέψεων για το 2011 καλύπτεται από τους πέντε αυτούς άξονες που προανέφερα με μια απόλυτη προτεραιότητα για τον πέμπτο άξονα που είναι ο άξονας των ανθρώπων. Αυτή η στρατηγική λοιπόν είναι στα τελευταία της στάδια για την πλήρη διατύπωσή της και ελπίζουμε ότι θα εγκριθεί ως ενούπο από το Συμβούλιο των Υπουργών. Δεν νομίζω ότι πρέπει να θεωρήσουμε όλοι ότι είναι υπόδειγμα και φάρος η Ισπανική κυβέρνηση, αλλά νομίζω ότι εν ταπεινοφροσύνη μπορούμε να παρουσιάσουμε αυτό το παράδειγμα της δράσης της Ισπανικής ε, ε, που θα μπορούσε να είναι ένα υπόδειγμα υλοποίησης αυτών των αρχών που έχουμε διακηρύξει σε ένα γενικό επίπεδο ως Προεδρία. Στη δεύτερη παρέμβαση ετέθηκε πάλι το θέμα της κοινωνικής διάστασης, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και μια αναφορά στην πρωτοβουλία GMS και σε θέματα όπου υπήρξε νομοθετική προσπάθεια από το Συμβούλιο. Αλλά ετέθη και το θέμα του ΙΤΕΡ, του Προγράμματος Θερμοπυρηνικής ε, Σύνδεξης. Σίγουρα η εμπιστοσύνη που τρέφεται προς το άτομό μου, όπως φαίνεται από το ερώτημά σας, θα απογοητευτείτε με το γεγονός ότι δεν μπορώ να σας δώσω μια πλήρη απάντηση υπήρχε η συμφωνία να εργαστούμε μέχρι την τελευταία στιγμή για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση για το πρόβλημα του ΙΤΕΡ που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό όπως το αναφέρατε. Έχει, είναι σαφής η διάγνωση και τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι τα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και η συμφωνία ήταν να δημιουργηθεί μια ομάδα εργασία. Και της οποίας ηγείται η Γενική Διευθυντής που είναι ε, στα αριστερά μου, που θα εργαστεί με το στόχο στις λίγες μέρες που μας έχουν μείνει να καταλήξουμε στη βέλτιστη πρόταση από την οποία θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αναζήτηση μιας λύσης. Εάν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα 100% τόσο το καλύτερο. Δεδομένης όμως της πολυπλοκότητας του προβλήματος δεδομένης της οικονομικής κατάστασης που διατρέχουμε. Και συμμερίζομαι απόλυτα αυτά τα οποία είπατε σήμερα το πρωί, δεδομένης της σημασίας αυτού του σχεδίου που είναι το πιο σημαντικό από τα πιο σημαντικά αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να βρούμε μια λύση βάσει της οποίας θα μπορέσουμε να έχουμε μια σύγκληση <clears throat> για να λυθεί τουλάχιστον ένα τμήμα του προβλήματος με τη συμμετοχή διαφόρων πηγών χρηματοδότησης. Δεν μπορώ να απαντήσω λοιπόν συγκεκριμένα σε ερωτήματα του αν θέλετε να ενταχθεί αυτό στο πρόγραμμα πλαίσιο, ομάδα από αυτό. Όχι, πρέπει να έχουμε μία ε, συνεργασία διαφόρων συνιστοσών από διάφορες κατευθύνσεις και αυτό είναι το πνεύμα μέσα στο οποίο δημιουργεί αυτή η ομάδα εργασίας που προανέφερα που δημιουργήθηκε μετά τη σύνοδο του, του, Υπουργικού, του Συμβουλίου Υπουργών Ανταγωνιστικότητας. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι όχι μόνο θάρρος, αλλά και ικανότητες εξέβρεση τη καλύτερη λύση, ώστε αυτό το σχέδιο να παραμείνει μέσα στα πλαίσια των αρχικών δεσμεύσεων και με τη βέλτιστη δυνατή λύση από οικονομική έποψη. Για την τρίτη παρέμβαση, που ήταν του κυρίου Λάγκε, αναφέρθηκε το θέμα των επενδύσεων για την καινοτομία ανεφέρθην προηγουμένως στο θέμα αυτό για την ισπανική εμπειρία, απαντώντας στην κυρία Ριέρα Μαδουρέντου, η ισπανική κυβέρνηση συνέταξε αυτή τη στρατηγική με τους πέντε αυτούς άξονες που έχουν σαν στόχο να ευνοήσουν τον επιχειρηματικό ιστό, να μην έχουμε μια προσέγγιση μονάχα ακαδημαϊκού χαρακτήρα, αλλά με την εμπλοκή και τη συμμετοχή των επιχειρηματιών Προσπαθήσαμε λοιπόν να φέρουμε στην πράξη τις αρχές αυτές που έχουμε διατυπώσει θεωρητικά και ελπίσουμε ότι θα έχουν την υποστήριξη και από το Συμβούλιο τον, το φθινόπωρο όταν τεθεί αυτό το σχέδιο για την καιροτομία. Τέταρτη παρέμβαση. Δεν ξέρω αν συμφωνούμε. Νομίζω ότι ήταν στην Γρανάδα, στην, στην συνάντηση της Γρανάδας, όπου είχε τεθεί ακριβώς αυτό το ερώτημα, όχι μόνο η κοινωνική διάσταση, αλλά και η εδαφική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνούμε ότι οι πολιτικές στα διάφορα επίπεδα διοίκησης, στα διάφορα εδαφικά επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι συμβατές μεταξύ τους. Και θέλουμε λοιπόν να είναι συμβατές και με την κοινωνική διάσταση και με την απαραίτητη προσοχή πρέπει να δοθεί στο εδαφικό επίπεδο. Όταν μιλάμε λοιπόν για την προώθηση και την υποστήριξη μηχανισμών απλοποίησης, γιατί έχουμε μιλήσει για την απλοποίηση, θεωρούμε ότι η απλοποίηση είναι και αυτή συμβατή με την προώθηση των συνεργειών μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων. Δεν πρόκειται μόνο για απλοποίηση των διαδικασιών, των υποβολών, προσκλήσεων κτλ. αλλά και μια γενικότερη συνέργεια μεταξύ των προγραμμάτων και με την συμβατοποίηση, όλο σα λέω τη λέξη συμβατοποίηση, αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την αρχή της αριστείας, η οποία είναι απαραίτητη για να υποστηριχθεί η κοινωνική συνοχή. Η αριστεία και η κοινωνική συνοχή θα πρέπει να είναι αμοιβαίως ε, συμβατές και να αλληλοενισχύονται ώστε τα προγράμματα και προσκλήσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος να αλληλοϊποστηρίζονται. Στη συνέχεια. Ο κύριος Βέβαια έλαβε το λόγο και με ρωτούσε σε ποιο βαθμό έχουμε προχωρήσει σε ό,τι αφορά τις, τα διπλώματα τεχνίες. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει ιδιαίτερα το θέμα αυτό στα Συμβούλια Ανταγωνιστικότητος, αλλά αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι θεωρούμε ότι η αλυσίδα δημιουργίας γνώσεως από την εκκίνηση της δημιουργίας της γνώσης δεν πρέπει πάντα να καταλήγει σε μια πρακτική εφαρμογή. Αφ' αυτής η έρευνα έχει αξία, αλλά θα πρέπει να δώσουμε και την πρέπουσα προσοχή στον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας της γνώσης, υποστηρίζοντας τις πολιτικές που έχουν να κάνουν με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Εν πάση περιπτώσει, είναι σαφές, και αυτό αναφέρθηκε στο Συμβούλιο ανταγωνιστικότητος ότι και οι υπουργοί βιομηχανίας έχουν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο για να αντιμετωπίσουν ακριβώς αυτή την πτυχή της έρευνας. Ο κύριος Τούρμες έκανε μια πολύ καλή σύνοψη της οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι χώρες μας και μέσα στο οποίο πλαίσιο χρειάστηκε να εργαστούμε και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο ΙΤΕΡ. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό έχει καλυφθεί από την απάντηση που έδωσα πριν από λίγα λεπτά. Έχω καλύψει λοιπόν το ζήτημα αυτό, πιστεύω. Για τον κύριο Έντσο, ανεφέρθη από αυτόν το θέμα του να μπορούμε να έχουμε μια πιο εύκολη δυνατότητα συμμετοχής σε όλα τα προγράμματα. Αυτό ήταν και ο στόχος της προσπάθειας μας για την απλοποίηση. Προσπαθούσαμε να διευκολύνουμε την, την πρόσβαση όλων στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δίνοντας ως το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και επίσης απλοποιώντας και τις διαδικασίες και το να μην έχουμε στεγανά προγράμματα τα οποία να είναι αποσυνδεδεμένα μεταξύ τους, αλλά με το να έχουμε συνέργεια μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων. Πιστεύω λοιπόν ότι σας έχω δώσει μια πρώτη απάντηση, κύριε Πρόεδρε, για όλα αυτά τα οποία συζητήθηκαν εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, για τις πληροφορίες ε, που μας δώσετε και σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για το ότι σε αυτούς τους έξι μήνες συνεργαστήκαμε τόσο καλά. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να διαβιβάσετε του χαιρετισμού μας και στην κυρία Υπουργό. Ήταν πολύ καλή η συνεργασία μας. Εύχομαι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τα ξαναλέμε εμείς εδώ πέρα στις 3 για την συνέχεια. Ευχαριστώ. Γεια σας.